Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε θερμά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, μια ακρόαση συγκεκριμένα, hearing. Ακρόαση λοιπόν για τη μεγάλη διάσκεψη του Ρίο του χρόνου στο Ρίο Ντεζανέρο της Βραζιλίας που Ρίο Συνήκωση, 20, έτσι αποκαλείται. Και σήμερα έχουμε εξαιρετικούς επαΐοντες υπό διαφορετικές ιδιότητες και αξιώματα που θα μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους και τις συστάσεις τους, οι απαιτήσει και εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε μια φιλόδοξη, ας το πω έτσι, ομάδα ένας όμιλος φιλόδοξων ανθρώπων που στα πιο διαφορετικά θέματα της αηφορίας στην ανάπτυξη τοποθετούμαστε και σε θέση με τους θεσμούς, στις ευρωπαϊκούς θεσμούς στις Βρυξέλλες είμαστε κινητήριος μοχλός κινητήρας. Το κάναμε αυτό και στη συζήτηση για την προστασία του κλίματος και για τη συζήτηση για τη βιοπικιλότητα και εμπλεκόμαστε σήμερα σε αυτό το θέμα. Ρίος είναι 20. Έχουμε εξαιρετικούς επαΐοντες τους χαιρετίζω όλους και τους καλωσορίζω. Πρωτού κάνουμε δύο γύρους. Πρώτο γύρο που εδώ στο Προεδρείο θα είμαστε και ο δεύτερος γύρος που βρίσκονται εν μέρη εδώ παρόντες και θα έρθουν εδώ πάνω στη συνέχεια, τον Άχιμ Στάινερ. Καλοχαιρετίζω πρώτα εκτελεστικό διευθυντή του προγράμματο για το περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών. Καλώς ήρθατε θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και στη συνέχεια Καρλ Φάλκενμπέργκ Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καρλ, καλώ όρισε θερμά. Χθε είμαστε από κοινού μαζί στην έναρξη τη πράσινη εβδομάδα. και γνωρίζουμε ότι στις 11 και 4 το πρέπει να αποχωρήσει σε άλλη, για άλλη εκδήλωση. Χαιρετίζω στο Προεδρείο τον Peter Gooders, senior economist, ε, οικονομολόγο, ανώτερο οικονομολόγο του ε, Ιδρύματος ε, της, για τη Διεθνή Ανάπτυξη. Καλώς ήρθατε και χαιρετώ εξ ευωνίμων την Μάρθα Χότσεβα Ρόχας από την Advocacy Care International. Καλώς ήρθατε κι εσείς παρόντες για το δεύτερο γύρο. Έχουμε τον Μπρίσλα Λόντ παρόντα, <clears throat> εκτελεστικό συντονιστή της, ε, Ευρω... Ε, Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Ρίο Συν 2012. Ε, Επίσης ο Ντέρεκ Όσμπον, πρόεδρος του Forum Stakeholders της Ουγγρικής Προεδρίας και στο, Ευρωπα... στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο τον Σάντορ Φίλεπ Καλώς ήρθατε. Αυτοί είναι οι παρόντες ήδη τώρα από το δεύτερο γύρο. Ο κύριος ε, ε, Νέιβα Ταβάρες θα έρθει υστερότερα στη συνέχεια. Χωρίς μεγάλες εισαγωγές και παρέμβαση είχα ήδη την ευκαιρία πρέπει να πω στην πρώτη διάσκεψη στη Στοχόλμη να είμαι παρόν και να παρακολουθήσω τα σχετικά πριν από 40 χρόνια Τότε υπήρχαν 3,8 δισεκατομμύρια κάτοικοι στην οικουμένη μας, στον πλανήτη μας. Άκουσα ότι τον Οκτώβριο εφέτος θα γεννηθεί <clears throat> εκείνος που θα συμπληρώσει το 7ο δισεκατομμύριο από πλευράς κατοίκων του πλανήτη. Και τι συμβαίνει σε εμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας σε κάθε οικογένεια από το πέμπτο παιδί κάνει ένα ειδικό δώρο Γίναμε λοιπόν πολλοί κάτοικοι του πλανήτη και τίθεται το ερώτημα ποια πορεία θα ακολουθήσουμε στο μέλλον εμείς ε, οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη Γη. Γι' αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Σας καλωσορίζω θερμά και δίνω αμέσως τον λόγο, αμέσως, στον εκτελεστικό διευθυντή, τον Άχιμ Στάινερ από τα Ηνωμένα Έθνη. Πέντε έως δέκα λεπτά ίσως στην παρέμβασή σας και μετά θα έχουμε και ερωτήσεις απαντήσεις ε, επόμενη παρέμβαση. Παρακαλώ, Αχιμ Στάινερ, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Τζο Λάνια. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, καλή σα μέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να σα προσφωνήσω εξ ονόματο των Ηνωμένων Εθνών και από κοινού με τον συνάδελφο Μπρίσλα Λόντ, επικεφαλή ε, του δεύτερου γύρου. Όπω είπε ο Γιώ όχι μόνο στρέφει το βλέμμα ο πλανήτη ε, στο Ρίο συν 20, αλλά και στην Στοχόλμη συν 40. Και τι προηγούμενε δεκαετίε ε, η διεθνή κοινότητα προσπαθεί να βρει και τα φόρα και τα υποδείγματα μέσα από τα οποία θα μπορεί να διαχειριστεί τον αυξανόμενο πληθυσμό του κόσμου που και την αυξανόμενη κατανάλωση διαρκώς με γεωμετρικούς ρυθμούς όλα και με τις περιβαλλοντικές αλλαγές που παρατηρούνται παγκόσμια είτε υπό την εθνική πτυχή και την πτυχή της ασφάλειας, την ενεργειακή ασφάλεια, επιστημιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των υδάτινων πόρων υπό οποιοδήποτε πρίσμα ή ε, τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, μια ξηρασία κάπου στον κόσμο μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις για την παραγωγή τροφίμων αλλού στον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι ζούμε σε περίοδο όπου η επιστημιστική ασφάλεια, η ασφάλεια τροφίμων, οι κλιματικές αλλαγές είναι θέματα που όλο και περισσότερο δεν είναι μόνο θέματα της διαχείρισης της περιβαλλοντικής διάστασης, αλλά ουσιαστικά της διαχείρισης ενός ευρύτερου φάσματος ε, για την ε, ανάπτυξη προς το μέλλον. Και όχι μόνο μόνο υπό το πρίσμα της αηφορίας, αλλά επίσης ε, και υπό το, το πρίσμα της ισότητας. Αηφορία και ισότητα, ισοδίκαια, ισοδίκαια ρύθμιση είναι νομίζω θεμελιώδη στοιχεία για το μέλλον των διεθνών σχέσεων καθοριστική σημασία. Αν δει κανεί παγκόσμια τον κόσμο σήμερα και τον γύρο των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο στην Τόχα, τι διαπραγματεύσει για το κλίμα, την αηφορία σε σχέση με τι ε, προτάσει ε, και στη Νέα Υόρκη, και όχι μόνο λόγω μιας διαφωνίας επί της ε, ουσίας, αλλά λόγω διαφωνιών για τις ε, κατεχόμενες ε, περιοχές, τότε μπορεί να κατανοήσει κανείς μια απογοήτευση όσον αφορά το πολυμερές πλαίσιο. Όχι μόνο ριζωμένη σε σχέση με κάποια στοιχεία αυτών των φόρων, αλλά όσον αφορά την διεθνή πολιτική, γεωπολιτική, πολιτική οικονομία, δράσεις για την ανάπτυξη. Από πλευρά ε, των ΗΕ να δημοσιοποιήθηκε μια έκθεση για την αποσύνδεση, decoupling, για την, ε, το Ίδρυμα για τους ε, διεθνείς πόρους, βλέποντας τους πόρους και την κατανάλωση τα επόμενα 40 χρόνια. Χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αυτή η έκθεση έχει προοπτικές σε τέσσερις διαστάσεις, ενέργεια, βιομάζα, άλλους φυσικούς πόρους, τριπλασιασμό συνολικά, συνολικά της κατανάλωσης των πόρων στις επόμενες δεκαετίες. Οποιοςδήποτε τώρα, είτε είναι οικονομολόγος, είτε είναι υπεύθυνο για πολιτικές στρατηγικές, είτε εμπλεκόμενος σε ένα πάνελ. Αυτό είναι ένα μη βιώσιμο σενάριο και είναι μια τεράστια πρόκληση. Και εδώ ερχόμαστε τώρα σε άλλη μια συνιστόσα, Ρίο συν 20 την αποκαλούμε. Ουσιαστικά το πνεύμα του Ρίο το 1992 όταν υπήρχε ένα επίπεδο συνένεσης τι πρέπει να γίνει σήμερα. Ξεκινώ όταν θα συνέλθουν στο Ρίο Ντεζανέρι τον Ιούνιο 2012, 20 χρόνια μετά το Ρίο, οι υπεύθυνοι σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό το οποίο θα βρεθεί είναι η αηφορία της ανάπτυξης εκείνοι που άρθρωσαν το όραμα ενός ε, υποδείγματος ως προτύπου, ενός ε, οδικού χάρτη προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να πορευθούμε, εκείνοι που στρέφουμε το βλέμμα στο Ρίο 2012 για να ξεκινήσουμε εκ νέου αυτή την πορεία, θα πρέπει να πω ότι η αηφορία στην ανάπτυξη εξακολουθεί να υφίσταται ε, και να αποτελεί στοιχείο εμπιστοσύνη όπως σήμερα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν καταφέραμε να επιταχύνουμε την ε, μετάβαση όσον αφορά την επίτευξη αυτού του υποδείγματος. Και εδώ ένα από τους στόχους της διάσκεψης, η αναθεώρηση όπως την αποκαλούμε και οι αναλύσεις γενικότερα για να κατανοήσουμε το τι έγινε και τι δεν έγινε για τους κινδύνους του, ε, της πολυμερούς αντιμετώπισης και της, ε, την, ε, τις κατηγορίες που εγείρονται πολλές φορές. Ε, κάποιοι λένε ότι δεν ακολουθείται ε, ταχεία πορεία σε σχέση για παράδειγμα με τις αναψιόμενες χώρες αλλά και όλους τους άλλους δείκτες και τα επιχειρήματα που έχουν αρθρωθεί. Στο κάτω-κάτω στόχος δεν είναι να δακτυλοδείξουμε τους υπευθύνους ή να εγείρουμε κατηγορίες αλλά να δούμε τα μαθήματα ποια είναι, γιατί δεν πορευθήκαμε αρκετά γρήγορα. Δεύτερον, στόχος θα είναι να δεσμευτούμε όσον αφορά και τις αρχές ε, της ε, ε, ημερήσιας διάταξης του 21ου αιώνα και σε σχέση και με την, το Ρίο 92, ε, όχι να ξανανοίξουμε κάποια θέματα, αλλά να υπάρξει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο πλαίσιο για μια ε, δημιουργική συζήτηση και αναζήτηση. Και όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται στο τραπέζι. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι οι κλιματικέ αλλαγέ είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά είναι και ένα αναδυόμενο, αναφιόμενο θέμα σε σχέση με τι σημερινέ γεωπολιτικέ πραγματικότητε. Βρισκόμαστε στην καρδιά πραγματικά πολύ δύσκολων κλιματικών διαδικασιών, όπου όσα συνέβησαν τα τελευταία 20 χρόνια ήταν μια εξαιρετική διαδικασία θέτοντας ένα θέμα από τη θεωρητική επιστήμη στο παρελθόν σήμερα σε μια πραγματική, ας το πω έτσι, σε μια πραγματικότητα, βλέποντας την ενεργειακή μας οικονομία, την κινητικότητα, το θέμα του να ενταχθούν αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, στην βιόσφαιρα, να προσαρμοστούμε σε σχέση και με το μέλλον της γεωργίας και όλα τα συναφή. Πιστεύω ότι βλέποντας το Ρίο, ιδιαίτερα από το πρίσμα, υπό το πρίσμα της Ευρώπης και υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι τιμή να είμαι εκπρόσωπος του, των Ηνωμένων Εθνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητώντας για το θέμα του τι σημαίνει ηγεσία, ηγετικό ρόλος σε μια χρονική συγκυρία που δεν έχει προετοιμαστεί ακόμα ο κόσμος ε, τέλεια για μια τέτοια διάσκεψη κορυφής. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου επουλώνουμε ακόμα τις πληγές μας παγκόσμια, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής, χρηματοοικονομικής παγκόσμιας κρίσης ε, και Είμαστε ως παγκόσμιοι παίκτες ε, στο παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει μια συνεκτική συναφής παγκοσμιοποιημένη ημερήσια διάταξη από κοινού μεταξύ όλων. Και υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα όσον αφορά τα αναπτυσσόμενα κράτη. Και για παράδειγμα δεν μπόρεσαν να ευθυγραμμίσουν τα συμφέροντά τους με τις μεγάλες οικονομίες οι αναπτυσσόμενες χώρες ήδη στην Κοπενχάγη και με τις διατλαντικές προοπτικές. Δεν υπάρχει μια σαφής ενιαία μόνη προοπτική για το μέλλον ως απάντηση την Ευρώπη για τις ε, διεθνείς πολιτικές για το κλίμα. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό λοιπόν και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα κοινό παγκόσμιο και οικονομικά εμπλεκόμενους ε, από τον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά, χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και την κοινωνία των πολιτών που προσβλέπει προς αυτή τη διεθνή κοινωνία, κοινότητα για να υπάρξει, να διασφαλιστεί αυτή η ηγεσία. Πολιτικά λοιπόν και τεράστιες προσδοκίες ότι το Ρίο συνήκωση θα μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία και να δώσει απαντήσεις για το πώς θα διαχειριστούμε τη μελλοντική μας ανάπτυξη στην οικουμένη, στον πλανήτη μας ε, ως ε, μια, ε, ένας πλανήτης με 7 δισεκατομμύρια εφέτος και 9 στο άμεσο μέλλον αν λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της, θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, διάσκεψης του χρόνου, πράσινη οικονομία, εκρίζωση της φτώχειας, θεσμικό πλαίσιο για την αηφορία στην ανάπτυξη, όλα αυτά αν τα δούμε. Έχουμε δύο θέματα που πραγματικά δεν ε, ανατρέχουν στα, στις θεμελιώδεις ε, αξίες της αηφορίας στην ανάπτυξη, αλλά το ερώτημα γιατί δεν κινηθήκαμε ταχύτερα, ποια μαθήματα πρέπει να συναγάγουμε. Κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη είναι σε τυχερή θέση, διότι μέσω της δικής της εξέλιξης ενός μιας ε, πολύ πραγμα... Ε, προοδευτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και το βλέπουμε αυτό και πώς ε, στις Βρυξέλλες και με τη δυναμική στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη κατάφεραν να αναβαθμίσουν αυτά τα θέματα και πολλές φορές κατάφεραν να, ε, το, να εντάξουν τις χώρες σε μια ταχύτερη πορεία, fast track, ε, σε σχέση με την προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθεια να κατανοήσουμε πώς αυτά τα μαθήματα σε σχέση με διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές προκλήσεις μπορούν ε, να διατυπωθούν αυτά τα μαθήματα. Στις πολλές συζητήσεις που είχατε ήδη στο πλαίσιο των κλιματικών, της πολιτικής για το κλίμα και για την βιοπικιλότητα και την Natura 2000 και την CAP, η αγροτική πολιτική και πολλά σε σχέση με τις ε, κατευθύνσεις για την εξέλιξη της ε, πράσινης οικονομίας. Επιτρέψτε μου να τονίσω εδώ τον τρόπο για τον οποίο εμείς ε, στα Ηνωμένα Έθνη αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα και ξεκινήσαμε να αρθρώνουμε με τις υπόλοιπες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ένα όραμα για την πράσινη οικονομία δεν είναι μία ακόμα πρόσθετα οικονομία. Αυτή η στρατηγική, αυτή η συζήτηση επικεντρώνεται στο πώς η σημερινή οικονομία θα μπορέσει να κινηθεί προς μια πιο πράσινη οικονομία που θα χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους πόρους, θα εκλεί λιγότερο άνθρακα και θα ε, υπάρχουν τα μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε σε σχέση με τις υποδομές να μην θεωρούνται απλά και μόνο μία ε, εκμετάλλευση πόρων αλλά αποκατάσταση και συντηρητική αποκατάσταση. Πολλά μαθήματα μπορούν να συναρθούν βλέποντας την πράσινη οικονομία. Πράγματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη εν μέρη ζείτε και βιώνετε και διαχειρίζεστε εσείς αυτά τα στοιχεία. Κινείται και ο βιομηχανοποιημένος κόσμος και υπάρχει και μεγάλη ταχύτητα. Είναι κάτι και που αφορά και τις αναδυόμενες οικονομίες. Η Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική ή άλλοι άλλοι που λένε κάποιοι ότι δεν προτίθενται να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να δούμε την οικονομική δομή τους και τις πολιτικές τους και σε σχέση με τη Βραζιλία και την Κίνα υπάρχουν σημαντικές μεταθέσεις. Υπό το πρίσμα των Ηνωμένων Εθνών δικό μας μέλημα είναι να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα 140 άλλα έθνη, αναπτυσσόμενες χώρες, ε, μικρές ε, χώρες και νησιωτικές χώρες ε, δεν θα βρίσκονται στο περιθώριο ή δεν θα μείνουν πίσω όσον αφορά την κοινή αυτή πορεία. Η διεθνής υποστήριξη για τις υποδομές βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής στο Ρίο και πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το εγχείρημα. Και για το άλλο τμήμα της συζήτησης δεν είναι συγκυριακό, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το πολυμερές σύστημα βρίσκεται υπό ενδελεχή εξέταση. Και βρισκόμαστε σήμερα στο επίκεντρο, στην καρδιά αυτών των θεμάτων. Ίσως στις Βρυξέλλες ε, μπορεί κανείς πιο ε, εύκολα και άμεσα να τα αντιμετωπίσει αυτά, να το πω με απλά λόγια. Ένα η πρότυπο για την αηφορία της ανάπτυξης δημιουργήθηκε και αρθρώθηκε στο Ρίο. Αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο μας καθυστέρησε. Με τρεις πυλώνες συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο με οικονομικά πρότυπα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Ουσιαστικά στο Ρίο θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την τριχοτομία, αυτή την ε, στεγανότητα μεταξύ αυτών των πυλώνων. Θα πρέπει να κινηθούμε σε μια κοινή τριπλή έλικα όπου να προσπαθήσουμε να συνενώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Η έννοια της ε, πράσινης οικονομίας είναι μια άρθρωση αυτού του λόγου, μια διατύπωση αυτών των επιχειρημάτων. Πρέπει περιβαλλοντικά, οικονομικά ε, και οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά να κινηθούμε σε ένα κοινό άξονα. Και αν δει κανεί ε, τις πολιτικές, η διασύνδεση είναι προφανή. Ο ΠΟΗ, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, εκτιμά ότι ένας στους 4, 25% θα πεθαίνουν πρόωρα λόγω της επιβάρυνσης των κλιματικών και περιβαλλοντικών, με συγχωρείτε, συνιστοσών πράσινες θέσει απασχόληση, μια νέα γενναία των οικονομική ανάπτυξη. Τι είδου ανάπτυξη στον σύγχρονο κόσμο θα έχουμε που θα επιτρέψει να αναπτύσσονται οι οικονομίε μα. Διότι κυρίε και κύριοι με νέα δι πληθυσμό πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται η παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την ανάπτυξη με βάση το πρότυπο του παρελθόντο. Ενώ θα ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο και θα αναθεωρούμε τη δομή των Ηνωμένων Έχουμε εδώ το θέμα της ε, διακυβέρνησης για τα θέματα του περιβάλλοντος. Αν πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο περιβάλλον και αυτά, αυτές θα είναι τόσο σημαντικές, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια παγκόσμια συνένεση, μια δυνατότητα να δράσουμε συλλογικά όλοι με δομές ε, για την ε, διακυβέρνηση που δεν θα είναι παροχημένες παλαιές ήδη προ 40 ετών, 4 δεκαετιών, αλλά θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα εγκρίνονται σε ένα άλλο

Φόρουμ, στη Γενική Συνέλευση. Και εκεί δεν υπάρχει με αυτό το πλαίσιο μια αποτελεσματική διακυβέρνηση για το περιβάλλον. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί η θεσμική δυνατότητα να μπορέσουμε από πλευρά ε, ε περιβάλλοντο να προσφέρουμε αυτό το οποίο ε, δημιουργήθηκε για τα θέματα υγεία. Ένα είδου ε, παγκόσμιο οργανισμό ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Άχιμ Στάινερ, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την πολύ έντονη, δυνατή εισαγωγή επιλογή με ένα σαφέστατο μήνυμα που μας δώσατε για την διάσκεψη Ρίο συν 20 και πραγματικά θα έπρεπε να είχαμε πει ότι θα έχουμε δύο ε, τμήματα πράσινη οικονομία πρώτο Πρώτα και διαχείριση, διακυβέρνηση της αηφορίας της ανάπτυξης. Δεύτερο τμήμα της ε, σημερινής μας, σημερινής μας ακρόασης. Εσείς στρέψατε το βλέμμα στο μέλλον και είπατε πώς μπορούν να ενισχυθούν τα θεσμικά θέματα και τα ιδρύματα, οι θεσμοί παγκόσμια και σε σχέση με την, ε, τον παραλυσμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και να είχαμε ένα Παγκόσμιο Οργανισμό για το περιβάλλον που θα μπορούσε με τέτοιες αρμοδιότητες και ταχύτητα να δράσει και να λαμβάνει αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν. Αηφορία στην ανάπτυξη. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη και είναι ένα μείζον θέμα αυτό μέσα στο πλαίσιο των ε, διασκέψεων των Ηνωμένων Θέλω να καλωσορίσω τον ε, Αντώνιο Βιτζιλάντε, εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών εδώ στις Βρυξέλλες, συνεργαζόμαστε σε σχέση με πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο. πρωτού δώσω τον λόγο τώρα στη συνέχεια στον Καρλ Φάρκενμπεργκ, Γενικό Διευθυντή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλωσορίζω τον Γιάρο Σλαβ Πέτρας, Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου. Τα 27 βλέπετε κράτη-μέλη και αυτά πρέπει να κάνουν στο Συμβούλιο τη δουλειά του ως ε, εμπλεκόμενοι σε σχέση και με εσάς τα, τα Ηνωμένα Έθνη. Καρλ Φάλκενμπεργκ λοιπόν για τις προσδοκίες όσον αφορά την Ευρώπη, ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την διάσκεψη. Ποια είναι τα κριτήρια, ο, ο γνώμονας, ο, ο πύχης που πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ για να σας και που παρουσιάσατε αυτό το ζήτημα τόσο ολοκληρωμένα. Και σε πολλά σημεία συμφωνούμε απόλυτα. Και μας μας ε, προβληματίζουν αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις τις οποίες αναφερθήκατε. υπάρχει προοπτική των 9 δισεκατομμυρίων κατοίκων μέχρι το 2050 και αυτή η δημογραφική ε, ανάπτυξη ε, διαδραματίζεται κυρίως στο αναπτυσσόμενο τμήμα ε, της Ιφιλίου. Συνεπώς, η αύξηση της ζήτησης θα είναι μεγαλύτερη από ότι αν η δημογραφική αλλαγή αυτή παρουσιαζόταν στο αναπτυγμένο ε, κομμάτι της υφηλίου. Μας προβληματίζουν οι επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι εξελίξεις σε επίπεδο φυσικών πόρων και στην Ευρώπη φέτος εστιάζουμε στην αποδοτικότητα των φυσικών πόρων. Πλέον ε, παίρνει το χαρακτήρα ε, προτεραιότητας για να διασφαλίσουμε ότι ότι θα μάθουμε το μάθημά μας, αν θέλετε, μέσα στην Ευρώπη και θα στρέψουμε τις οικονομίες μας ε, προς ε, μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε επίπεδο πόρων, ε, απομάκρυνση από την ηλική διάσταση όσο αυτό είναι δυνατό και να εστιάσουμε και στην οικονομία της ανακύκλωσης από ό,τι της κατανάλωσης και απόρριψης. Μας απασχολούν λοιπόν όλα αυτά τα παγκόσμια φαινόμενα και ανυπομονούμε κι εμεί ε, να πάμε σε αυτή τη διάσκεψη στο Ρίο Συνήκωση. Η Επιτροπή οριστικοποιεί τώρα μία ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που θα περιλαμβάνει ε, τη δική μας οπτική γωνία για την διάσκεψη αυτή και για τα πιθανά αποτελέσματα. μετά από μακροσκελείς συζητήσει με κύριο θέμα την πράσινη οικονομία ως όχημα προς ε, την βιώσιμη ανάπτυξη και το ζήτημα της ε, διακυβέρνησης που αναφέρθηκε προηγουμένως. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες, πολλές ευκαιρίες, αλλά και ε, πολλά εμπόδια να επιπηδήσουμε. Νομίζω ότι η παρουσίαση του κυρίου Στάινερ ήταν σαφής και αντικειμενική. Ε, το θέμα δεν είναι ότι δεν κατανοούμε τις προκλήσεις. Η πρόκληση στο ορίο συνήκωση θα είναι να αναπτύξουμε, να ε, κατανοήσουμε από κοινού ε, το τι συμβαίνει ε, και να συμφωνήσουμε στα προβλήματα αντί να κοιτάμε τι μπορεί να κάνει η άλλη πλευρά. Τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και επί της ουσίας πολλά ακόμα μένουν να γίνουν. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο τι πιστεύουμε ότι θα συμπεριλαμβάνει μια πράσινη οικονομία. Να επικεντρωθούμε στο ποιος κάνει τι και προς ποια κατεύθυνση. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της πράσινης οικονομίας. Όπως είπα θα πρέπει να υποστηρίζει την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή Ε, να ευθυγραμμίζει κατά κάποιο τρόπο τις ε, ε, προσδοκίες μας σε επίπεδο ζωής, σε επίπεδο ποιότητας ζωής, με τις αντικειμενικές συνθήκες σε επίπεδο περιβάλλοντος και τους περιορισμούς που μας περιλαμβάνει. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι στο ότι αυτό δεν αφορά μόνο τις ε, διάφορες επιτροπές ε, περιβάλλοντος. Αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και την, τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και δυνατότητες και να εξηγήσουμε σε όλο τον πληθυσμό της οικουμένης ότι η οικονομία ότι η πράσινη οικονομία μάλλον δεν θα εμποδίσει ε, την ε, πραγματική οικονομία, αλλά θα τη βοηθήσει να εξελιχθεί περαιτέρω. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε πολύ συγκεκριμένα τι εννοούμε με τον όρο πράσινη οικονομία, τι μπορούμε να περιμένουμε από το Ρίο Συνήκωση, ε, με την επένδυση σε πόρους και φυσικό κεφάλαιο, να κατανοήσουμε ότι το φυσικό κεφάλαιο αναφέρεται σε πολύ ε, σημαντικούς πόρους όπως το νερό και τα λοιπά. Ε, να εστιάσουμε στην ανακύκλωση των αποβλήτων και ούτω καθεξής. Αν οδεύσουμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση, οι κύριες μελέτες ε, εξηγούν γιατί αυτές υπηρεσίες οικοσυστημάτων <clears throat> πράσινης οικονομίας είναι, είναι πολύ σημαντικές στις ε, αρμόδιες χώρες. Γιατί προς το παρόν οι χώρες αυτές δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να έχουν δικές τους εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού ε, που παράγει και πάλι καθαρό νερό. καθαρό νερό για πάνω από τέσσερα δις ε, κατοίκους αυτής της γης. Αυτό το νερό λοιπόν παράγεται ακόμα από τη μητέρα φύση και αν δεν έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να παράξουν αυτό το νερό, δεν θα έχουν νερό. Πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα. Να τα κατανοήσουμε όλοι πολύ καλά, μετά να συζητήσουμε για το ποιες είναι οι παράμετροι, οι ενδείξεις που μπορούμε να εισαγάγουμε στην οικονομία, ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς ε, να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση αυτών των περιορισμών. Θα μιλήσουμε για την κοστολόγηση, συστήματα φορολόγησης. Ακόμα με εκπλήσει όταν σε πολλές πολλές χώρες του κόσμου βλέπω ότι υπάρχει ακόμα φόρος ε, στην απασχόληση αντί να φορολογούμε τις ε, πραγματικά ε, σπάνιες πρώτες ύλες, τους φυσικούς πόρους. Τα συστήματά μας έχουν τη δυνατότητα να καταστούν πλήρως παραγωγικά, αλλά αν φορολογούμε τους λάθος πόρους, δηλαδή την απασχόληση, τότε δεν μπορεί να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ε, οι ευκαιρίες για απασχόληση όλο ένα και μειώνονται ενώ αυξάνεται η παραγωγικότητα. Και δεν φορολογούμε τους ε, φυσικούς πόρους που είναι και σπάνιοι. Κάτι άλλο στο οποίο θα πρέπει να στοχεύσουμε είναι οι φορείς και οι διάφοροι παράγοντες. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο όπου οι κυβερνήσεις ε, συζητούν στο Ρίο. Πρέπει να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές αρχές, πόλεις, ε, ενώσεις αγροτών. Όλοι αυτοί πρέπει να έλθουν στο Ρίο, να συζητήσουν και στο τέλος να αποδεχθούν ε, να δουλέψουν από κοινού προς μια κοινή κατεύθυνση. Βεβαίως και υπάρχουν δυσκολίες και παγίδες, γιατί όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη ατζέντα υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Ελπίζω να μην ε, καθίσουμε για πολύ καιρό να σκεφτούμε τι μαθήματα μπορούμε να αντιλήσουμε από το παρελθόν. Το Ρίο Συνήκο θα πρέπει να έχει το βλέμμα στραμμένο προ το μέλλον και όχι προ το παρελθόν. Στα διάφορα διεθνή φόρα, αυτό έχουμε κάνει κατά κύριο λόγο. Ε, ε, εστιάσαμε στο παρελθόν γιατί κάναμε αυτό και όχι το άλλο, γιατί δεν κάναμε αρκετά. Αλλά μπορούμε να χάσουμε πολύτιμο χρόνο συνεχίζοντας αυτό το εγχείρημα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα προς το μέλλον να προσδιορίσουμε τους στόχους μας βάσει ε, του επίπεδου ανάπτυξής μας. Ε, η Ευρώπη είναι ο καταξοχήν ε, πολυμερής ε, εταίρος γιατί απαρτίζεται έτσι κι από πολλά μέρη. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε και τους υπολείπους αλλά και ο θεσμός ο οποίος θα ιδρυθεί από εκεί θα είναι κάτι που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, ε, σοβαρή συζήτηση στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη δεν χτίστηκε, δεν οικοδομήθηκε μέσω της ομοφωνίας. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες βρήκαμε τον τρόπο να καταλήξουμε σε συμφωνίες με την ομοφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή ε, προετοιμάζει μια ανακοίνωση, πολύ καλό αυτό, και εμείς ε, στο Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο θα την εξετάσει την ανακοίνωση αυτή μάλλον μετά το καλοκαίρι και θα δούμε πώς ε, μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο συντονισμός μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Θα συνεχίσω τη συζήτηση με τον Πίτερ Βούντερς, ε, ανώτερο οικονομολόγο ε, της σχολής, ε, του Ιδρύματος Περιβαλλοντικών Εξελίξεων. Βεβαίως και είναι ο πλέον Δήμο να μας απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Να αναφερθώ σε κάποιες από τις δράσεις οι οποίες μπορεί να αναλυφθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε για το, άνω, το ποσοστό άνω του 20%. Να επανέλθω στις εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με το τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει στα πλαίσια στρατηγικής του 2020. Αν κοιτάξει όμως καταρχάς κανείς το θέμα της πράσινης οικονομίας, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πετύχει κανείς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι εθνικές αντιλήψεις, οι εθνικές συνθήκες, απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις, βελτιώσεις των συστημάτων, σωστές εφαρμογές, νέες διεθνείς συμφωνίες. Τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πράσινη οικονομία. Στα πλαίσια της προοπτικής του ερευνητικού μας προγράμματος είπαμε ότι η εναλλακτική λύση είναι το business as usual. Το business as usual είναι μια επιλογή που έχει κόστος και το κόστος αυτό πλέον δεν είναι Συνεπώς λοιπόν ας προσπαθήσουμε να περάσουμε σε μια διαφορετική ε, ε, αντίληψη. Ήμουν συγγραφέα σε ένα από, τα πρώτα, από τις πρώτες εκθέσεις για την πράσινη οικονομία ε, Νομίζω ότι ο κύριος Φάλκεμπεργκ σας εξήγησε πολύ καλά ότι αυτό που χρειαζόμαστε στην οικονομία είναι τα κίνητρα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη το τι πράγματι είναι η πράσινη οικονομία. Αυτό είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να περάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε πράσινη οικονομία. Το θέμα είναι με ποιες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε εντοπίσει κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο χωρίς ε, να υπάρχει ανάγκη περίπλοκων ε, συμφωνιών διεθνών και προστατεύοντας τα συμφέροντα των ε, διαφόρων κρατών. Θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία η οποία να βοηθά να ληφθούν τα μέτρα αυτά και θα πρέπει και τα συστήματα αυτά Φαίνεται ότι υπάρχουν μερικές φορές ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα αυτό και ελπίζουμε ότι το σύστημα της πράσινης φορολογίας είναι κάτι το οποίο σε κάποια στιγμή εν πάση περιπτώσει θα εξαπλωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και συστήματα και συμφωνίες οι οποίες είναι σχετικά αντίθετες με αυτό το οποίο εννοούμε πράσινη οικονομία. Ε, πρέπει να ξεκινήσουμε με τέτοιο τρόπο υπολογισμού των μέτρων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε οι οικονομίες να γίνουν πιο αηφόρες. Η οργάνωσή μου έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία η οποία ονομάζεται Global Subsidies Initiative. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τα ορυκτά καύσιμα. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ υψηλό κόστος, 700 δις κατέτος, το 1% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν ενισχύσουμε την οικονομία. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει σε σχέση, εν περιπτώσει, ε, στον τομέα των επιδοτήσεων είναι το να δει κανείς πόσο λίγα γνωρίζουμε γύρω από αυτό το θέμα. Έχουν γίνει προτάσεις προς την ε, ομάδα των 20. Η ομάδα των 20 έχει αντιμετωπίσει το θέμα των επιδοτήσεων Νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των ε, σκέψεων αυτών αν ε, δεν αντιμετωπίσουμε τα άσχημα παραδείγματα τα οποία μερικές φορές ε, οι ίδιοι δίδουμε. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και με αντίθετες με την έννοια των επιδοτήσεων αποφάσεις όπως το θέμα της απαλλαγής φορολογίας μερικές φορές για ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, τα καύσιμα αυτό είναι κάτι το οποίο στην ουσία είναι να μην ενθαρρύνουμε ε, κάποια μέτρα τα οποία θα έπρεπε να προωθούμε αντίθετα. Ε, κάποιοι βέβαια λέγουν ότι τέτοιου είδους μέτρα είναι κίνητρα, κίνητρα απαραίτητα, αλλά η απόφαση η οποία έχει ληφθεί στις περισσότερες χώρες είναι η επιλογή της αύξησης της παραγωγής και συνεχούς αύξησης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Διαρωτώ με αυτό θα μας βοηθήσει στο μέλλον ή θα μας αγκυρώσει σε ένα μέλλον το οποίο θα μας βρει πλήρως εξαρτημένος από την οικονομία των ε, υδρογών ανθράκων. Νομίζω ότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από αντιπαραγωγικές ενέργειες τις οποίες δυστυχώς συνεχίζουμε να προβαίνουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν επίσης και οι αγορές γενικότερα και στον τομέα των υπηρεσιών και στον τομέα των ε, αγαθών και φυσικά είναι ένας τομέας οι αγορές ε, στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτιδα θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο και στον τομέα των δημοσίων προμηθειών και στον τομέα των συνεργειών ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και όταν ε, εξετάζει κανείς αυτές τις εταιρικές σχέσεις, βλέπει ότι τα κριτήρια τα περιβαλλοντικά τα οποία περιλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές τις εταιρικέ είναι ελάχιστα τις περισσότερες φορές και δεν λαμβάνονται σοβαρά, σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει βέβαια και έχει πάρει κάποια μέτρα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε έναν άλλο τομέα, ο οποίος είναι θα έλεγα γενικότερα εμπόδιο, αλλά μπορεί να γίνει και ευκαιρία. Είναι οι βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν με εντατικό τρόπο την ενέργεια. Αν δείτε τις ιστοσελίδες οργανώσεων, όπως η παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου, η χάλιβα, θα δείτε ότι υπογραμμίζουν τον ρόλο που μπορούν τα προϊόντα τους να παίξουν στα πλαίσια μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας η οποία παράγει λιγότερες εκπομπές. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τις μεταφορές στον τομέα των αυτοκινήτων, στον τομέα των μηχανισμών που απαιτούνται και των εξοπλισμών των τεχνικών που απαιτούνται για την ε, οικονομικότερη και αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας. Πιστεύουν λοιπόν οι βιομηχανίες αυτές ότι μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα της, ε, της ε, μιας οικονομίας περισσότερο πράσινη, θέλουν να πάρουν μέρος στην επεξεργασία τομέων στους οποίους μπορούμε να χαμηλώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Είναι ένας τομέας νομίζω νέος σχετικά σε συνεργασία με αυτές τις βιομηχανίες και ε, τελικά όμως η οικονομία είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει τις καλύτερες, την έβρεση και την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων. Φοβάμαι ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν για επενδύσεις στον τομέα του πρασινίσματος της οικονομίας δεν είναι οι καλύτερες. Πρέπει τουλάχιστον να, γίνουν εξίσου καλές με τις υπόλοιπες επενδυτικές δυνατότητες σε παραδοσιακούς τομείς. Ε, συνεργαζόμαστε και με τον ΠΟΕ και πολλές φορές οι αποφάσεις δεν είναι πάντα θετικές. Εμείς στη Διεθνή Οργάνωση για την Αϊφόρο Ανάπτυξη πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν ορισμένες πιλωτικές πρωτοβουλίες υψηλής θα έλεγα επίπτωσης και επιρροής. Ε, θα μπορούσαν χώρες να πούν ότι θα αφαιρέσουν όλες τις επιδοτήσεις στην κατανάλωση ενέργειας εφόσον δεν είναι θετικές για τη μείωση της κατανάλωσης ή δεν είναι υπέρ <coughs> της, της παραγωγής ενέργειας από πράσινες πηγές. Τότε θα περάσουμε το στόχο του ποσοστού 20% με εναλλακτικούς βέβαια πάντα στόχους. Το θέμα του τμήματος, του κατεχόμενου τμήματος της αγοράς ε, προκαλεί πάρα πολλές συζητήσεις και σε επίπεδο πάνελ του ΠΟΕ με την Κίνα. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το τίμημα για να γίνει πολιτικά αποδεκτή η αντίληψη αυτή. Οι συμφωνίες αυτές δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι επίσημες διεθνείς συμβάσεις ή θα είναι ανεπίσημες σε επίπεδο συμφωνίας κυρίων έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε χρήση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουμε επίσης να προχωρήσουν οι συζητήσεις και με τις βιομηχανίες υψηλής εντατικής κατανάλωσης ενέργειας, να δούμε τι ακριβώς είναι οι ανάγκες που έχουμε σε επίπεδο CCS καθ' όλη τη διάρκεια ζωής αυτών των εγκαταστάσεων και να συζητήσουμε επίσης και το θέμα της ανταγωνιστικότητας με το καλύτερο δυνατό τρόπο. από ένα think tank, το Policy Research Institute, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει ηγετική θέση εφόσον είμαστε πεπισμένοι μόνο ότι η πράσινη οικονομία είναι το μέλλον. Yeah, Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ, Πέτρο Γκούντας. Η ομάδα προβληματισμού Think Tank έχει σκεφτεί, έχει αναλύσει, υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις που είναι πολύ καλές και για την ε, δημοσιονομική πολιτική και την ε, οικονομική πολιτική που πρέπει να εξετάζεται ως προς την αηφορία της. Οι Υπουργοί Οικονομικών είναι οι αγιατολάδες του παλαιού συστήματος που παραμένουν σε παλές δομές ε, προσκολλημένοι και είναι σχετικά συντηρητικοί και θα έλεγα το πράσινο κίνημα πρέπει και αυτό να φτάσει και αυτό στα κονδύλια τα δημοσιονομικά διότι με την οικονομική, τον οικονομικό αναπροσανατολισμό μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θετικές ιδέες που τις σημειώσαμε. Περνάμε στη συνέχεια στην επόμενη εισήγηση. Μάρτα Χουτσένα Ρόχας που ήταν επανειλημμένα είχε δραστηριοποιηθεί για αυτά τα θέματα στο παρελθόν παλαιότερα στην UCN, τώρα σήμερα στην Care International. Προσδοκούμε να ακούσουμε τις δικές σας παρατηρήσεις. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να παρευρεθώ εδώ σήμερα και να συμμετάσχω στη συζήτηση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την ανανέωση της πολιτικής δέσμευσης για την εξέβριση ενός ε, προγράμματος δράσης που προσανατολίζεται στις δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κύρια ευθύνη ε, να δώσει το καλό παράδειγμα της ε, μιας οικονομίας χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλά και θα δώσει ένα πρότυπο, ούτω ώστε οι αναπτυσσόμενες ε, χώρες να ακολουθήσουν ε, την ίδια οδό. Ακούσαμε μία από τις δυσκολίες που παρατηρείται μέχρι ε, τώρα, ότι δηλαδή λειτουργούμε με στεγανά. Εγώ θα πάω λίγο παραπέρα. Το κύριο πρόβλημα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ότι μένει εντός του τομέα του περιβαλλοντικού. Πολλέ από τι προσπάθειες που έχουν ε, καταβληθεί λοιπόν ε, στον τομέα αυτό περιορίζονται ε, σε, στην περιβαλλοντική διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά και για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και στις δύο ατζέντε αυτό το πρόβλημα. Η πράσινη οικονομία μας δίνει πολλά εργαλεία όμως για να ε, συνδυάσουμε την οικονομία και το περιβάλλον. Πολλά έχουν γίνει σε αυτό το πεδίο. Θα πρέπει όμως να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, διάσταση της ισότητας, equity, ε, στην πράσινη οικονομία. Εκεί θα εστιάσω εγώ σήμερα. Δηλαδή, πράσινη οικονομία αλλά και εξάλληψη, εκρίζωση της φτώχειας. Η δική μου οργάνωση προσπαθεί να καταπολεμήσει τη φτώχεια εδώ και 60 χρόνια σε 70 χώρες. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, εξετάζοντας την πράσινη οικονομία με ενόψη του Ρίο, προτεραιότητα είναι ε, να εξετάσουμε την σημασία της εξάλληψης της φτώχειας. Πολλέ προσπάθειες έχουν καταβληθεί βέβαια, αλλά βλέπουμε πάνω από ένα δις ε, ανθρώπου που, που ζουν υπό καθεστώ ακραίας φτώχειας και υποφέρουν από ε, την πείνα. Αυτό αποτελεί λοιπόν μία από τις κυριότερες προκλήσεις. Επομένως είναι σημαντικό, ε, καθώ η Ευρώπη οδεύει προ το Ρίο, η προτεραιότητα της εξάλληψη τη φτώχεια να βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα μα αλλά και για την ε, δημιουργία της, ε, και ανάπτυξη της ιδέας της πράσινης οικονομίας. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ε, ότι υπάρχει ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο των γυναικών τόσο στην πράσινη οικονομία όσο και στο ορίο συνήκωση. 70% των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι γυναίκες. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτες οι γυναίκες στις κλιματολογικές αλλαγές, αλλά δεν είναι μόνο θύματα, είναι και φορείς ε, αλλαγής. Γιατί παράγουν ε, τροφή, ε, προσφέρουν μάλλον τροφή, νερό, και πρώτε ύλε στι οικογένειέ του σε όλο τον κόσμο. 60 με 80% τη τροφή παρέχεται από τι γυναίκε. Σίγουρα θα έχετε ακούσει τέτοιε περιπτώσει. Ταυτόχρονα όμω, ακόμα και αν οι γυναίκε είναι υπεύθυνε για τη διαχείριση των πόρων, τη βάση δηλαδή τη πράσινη οικονομία, και ε, έχουν πνεύμα καινοτομία, δεν έχουμε ε, ε, αφιερώσει αρκετή προσοχή στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για ε, το Περιβάλλον για το Μάρτιο του 2010, είναι σημαντικό να τονίσουμε τον ηγετρικό ρόλο που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη του Ρίο Συνήκωση. Τρίτον, θα ήταν χρήσιμο όπως έχει ήδη προταθεί, να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για τον τομέα της ενέργειας, γιατί βεβαίως και η κλιματική αλλαγή είναι κύριο ε, σημείο και θα πρέπει να συμμετάσχει ε, ο τομέας της ενέργειας. Αλλά επίσης και η επιστηστική ασφάλεια και η γεωργία είναι τομείς που θα πρέπει να συμμετάσχουν ε, γιατί επηρεάζουν ε, τις διάφορες κοινωνικο-οικονομικές ε, πτυχές της πράσινης οικονομίας. 75% του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτάται από την γεωργία. Η φτωχή συνεχώς εκτίθεται παραπάνω σε χαμηλά επίπεδα, σε υψηλά επίπεδα ανασφάλειας επιστηστικής. ε, έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον θα έχουμε ένα πληθυσμό 9 δις ανθρώπων μέχρι το 2050. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Γιατί εκτιμάται ότι πρέπει να αυξηθεί κατά 70% η παραγωγή δηλαδή, χωρίς να καταστρέψουμε τον πλανήτη βεβαίως. Ταυτόχρονα, ένα τρίτο το, της παραγόμενης τροφής ε, πετιέται στα σκουπίδια. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς ε, θα βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της ε, ε, προσφοράς και της ζήτησης, αλλά και να καταρρύψουμε τα σταγανά. Να δούμε για παράδειγμα τις επιπτώσεις της πτυτικότητας των τιμών. Ε, θα μπορούσε λοιπόν να μας βοηθήσει αυτή η δυνατότητα να ενισχύσουμε περισσότερο αυτή την ιδέα της πράσινης οικονομίας. Θα ήθελα να πω εδώ, είναι σημαντικό το EU ε, Green Paper, η πράσινη Βιολογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, για να έχουμε μια νέα προσέγγιση προς τις περιβαλλοντικές πολιτικές. σε τελευταία ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αναφέρθηκε και αυτό το σημείο. Τέταρτον, ε, προϋποθέσεις ενίσχυσης ε, προσπαθειών. Δεν θέλω να, να δείξω κάτι με το δάχτυλο, αλλά ξέρουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται ένα τέτοιο πλαίσιο που θα τις ενισχύει και χρειάζονται και δημοσιονομικούς πόρους. Δύο σημεία θα ήθελα να τονίσω από αυτή την πλευρά. Πρώτον, βεβαίω, οι αναπτυσσόμενε χώρε θα πρέπει να επιτύχουν τις δεσμεύσεις Ε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος ε, δωρητή, αλλά πέρσι μόνο εννέα χώρες πληρούσαν τα κριτήρια και του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ανάγκη να το συμπληρώσουμε, συμπληρώσουμε αυτή τη χρηματοδότηση με εταιρικέ σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αλλά και να ε, καλύψουμε τις ανάγκες, ε, ε, τις ανάγκες αυτών που τις χρειάζονται περισσότερο. Επενδύσεις στην πράσινη οικονομία. Αυτό περιλαμβάνεται και στην πράσινη βίβλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει Ε, να μας σταματήσετε να διασφαλίζουμε ότι οι φτωχοί έχουν πρόσβαση στην τροφή, στο νερό, στην ε, υγεία, υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση κτλ. Όχι μόνο η ποσότητα της ενίσχυσης, αλλά και η ποιότητα της ενίσχυσης είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή όλες αυτές οι ενισχύσεις θα πρέπει να έχουν ε, σωστούς ε, μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητάς τους. Τα αποτελέσματα λοιπόν του 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνουν και αυτό το πλαίσιο ενδυνάμωσης και ενίσχυσης. Τέλος, για την υπευθυνότητα. θα ήθελα να τονίσω μία πτυχή αυτού του ζητήματος που δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ. Αντιλείται και από το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων για το πόσο δηλαδή είναι υπόλογες αυτές οι οργανώσεις προς τους δωρητές τους. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε ε, τα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουν, ε, το ώστε οι επενδύσεις που κάνουμε στην πράσινη οικονομία έχουν θετικές επιπτώσεις στην εξάλληψη της ε, φτώχειας. Εδώ θα ήθελα λοιπόν ε, κλείνοντας να πω ότι περιμένουμε πολλά, έχουμε μεγάλες προσδοκίες από το Ρίο 2020, στην 20 μάλλον. Ε, και ελπίζουμε να συμβάλλει στην εξάλληψη της φτώχειας. Ευχαριστώ. Thank you very much, ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρόφας. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η παρουσίασή σα, δηλαδή ε, η βιωσιμότητα έχει τρεις, βασίζεται σε τρει πυλώνε και όχι μόνο σε έναν. Εμείς βεβαίω, εστιάζουμε περισσότερο στην οικολογική πτυχή. Ελπίζω και συνάδελφοι από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να θα ε, ε, κάνουν την ίδια ακρόαση. Βεβαίω και όλα αυτά συνδέονται άμεσα με τι επενδύσει. Σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε για τα MDGs αλλά και για τον ρόλο των γυναικών, ιδιαίτερα στι αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε 10 λεπτά αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε τέσσερις που έχουν ήδη ζητήσει τον λόγο. Ένα λεπτό έχουμε συνηθίσει στις παρεμβάσεις. Θα καταφέρουμε μόνο αν ε, ο καθένας επί ένα λεπτό παρεμβαίνει να έχουμε σύντομες απαντήσεις γιατί θέλουμε να έχουμε αρκετό χρόνο για το δεύτερο γύρο, τη δεύτερη φάση στις και τέταρτο. Ρίχαρτ Ζέμπερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους εισηγητές για τις εξαιρετικές ε, εισαγωγές που μας έδωσαν στο θέμα και, και ακούσαμε. Δύο έννοιες ε, έχουν ρόλο κλειδιού θα έλεγα προώθηση των γυναικών. Οι γυναίκες είναι η ραχοκοκαλιά κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και εδώ θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν ό,τι περνούν από το χέρι τους για να βοηθήσουν να προωθούν οι γυναίκες. Δεύτερον, η αυτο ε, η υπεύθυνη θέση και δράση, ιδιαίτερα σε σχέση με την επικέντρωση των μικρών προγραμμάτων. Όσο μεγαλύτερα είναι τα προγράμματα, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κονδύλια και περισσότερα και εμπλοκή των κρατών. Και έτσι δεν είναι η σωστότερη χρήση των κονδυλίων, ιδιαίτερα στα μικρά, ε, μικρής εμβέλειας προγράμματα. Και ο ρόλος ε, των ε, γεωργιών για την food security, την επισητιστική ασφάλεια και οι περιβαλλοντικοί στόχοι αυτόματα θα επιτευχθούν αν έχουν την ευθύνη που θα αναλαμβάνουν οι γυναίκες και έχουμε και αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης. Ένα λεπτό τέλεια. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Κάνουμε λόγο για την πράσινη οικονομία σαν να είναι μια υποοικονομία ως υποκατηγορία. Λάθος ο τρόπος αντιμετώπισης αυτός των πραγματικών προκλήσεων για να μπορέσει η οικονομία που έχει δεσπόζοντα ρόλο στον πλανήτη μας να, πρέπει να γίνει πιο πράσινη. Θα ήθελα να αποφύγουμε και τον όρο πράσινη. Να γίνει πιο αποτελεσματική θα ήταν το σωστότερο. Λέγοντας πράσινη θέτουμε στην οικολογική γωνιά τα πράγματα. Στριμώχνονται εκεί. Θα ήθελα να πω αυτό που είπε ο Μπιλ Κλίντον. Η οικονομία είναι χαζούλη. Αυτή τα ρυθμίζει όλα. Πρέπει να είναι λοιπόν πολύ πιο αποτελεσματική με τις νέες ρυθμίσεις και προσαρμογές η οικονομία. Αποτελεσματικότητα και υψηλές τιμές των πόρων είναι καλή υπόθεση και θα μας κάνουν όλα αυτά πιο αποτελεσματικούς. Ερώτησή μου, Μπορούμε να τα συζητάμε αυτά επί ιστοδιεινεκές μεταξύ κυβερνήσεων. Η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι πώς θα εμπλακούν οι επιχειρήσεις ώστε να μπορέσει αυτός ο στόχος να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Margaret Όκ, παρακαλώ. Θα μπορούσα να συνεχίσω απόλυτα να γίνουν τα πράγματα πιο αποτελεσματικά. Να χρησιμοποιούμε τον όρο πράσινο ή οποιονδήποτε άλλο ρόλο. Αλλά σε σχέση με τα όσα αντιμετωπίζουμε, η πραγματική πρόκληση είναι δεν είδαμε κανένα πρότυπο ή παράδειγμα τα τελευταία 40 χρόνια από τη Στοχόλμη το 1972 για μια οικονομία, για την αποσύνδεση σε σχέση με τα θέματα ανάπτυξης, ακόμα και με παραδείγματα στη Δανία, στον ενεργειακό τομέα. Αυτό έγινε επειδή εισάγαμε αυτή την ε, νέα προσέγγιση. Ξέρω ότι είναι μια παλιά συζήτηση αυτή, αλλά αυτή η παλαιά συζήτηση για αυτά τα θέματα αναφέρει ήδη πριν από πολύ καιρό ότι πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους. Βλέπουμε ότι αυξάνεται ο λοιμός, η πείνα στον κόσμο, τα προβλήματα αυξάνονται και κανένας δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα και αυτές τις προκλήσεις. Ότι η οικονομία δεν επαρκεί αν δεν υπάρχει πραγματική αηφορία που ποτέ δεν είδαμε να υπάρχει μέχρι σήμερα. Τα ακούμε σε σχέση με ε, το επιζητούμενο αλλά δεν γίνεται πράξη. Γιατί αυτό το θέμα δεν τίθεται στο τραπέζι. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε στα κράτη-μέλη το θέτουν στο τραπέζι. Και στη δική μου τη χώρα, στη Δανία και στους πράσινους αριστερούς στη Δανία, δεν το θέτουμε στο τραπέζι, δεν το αντιμετωπίζουμε για να επιληθεί όπως πρέπει. Και αν δεν το κάνουμε αυτό θα καούμε. Ευχαριστώ. Καλ, εσείς τι θα λέγατε. Μία ερώτηση θα είχα εγώ. Ναι, εσείς παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες. Βρισκόμαστε σε πολύ ε, δύσκολες ε, συγκυρίες όσον αφορά την πολιτική και τα προβλήματα και τις προκλήσεις και ο λαϊκισμός ε, ε, βρίσκεται στην ανιούσα στην Ευρώπη και πραγματικά είναι σημαντικό να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση από τους υψηλά εμπλεκόμενους. Σε αυτό το σημείο θα είχα ένα σχόλιο, κάθετο ερώτηση, σχόλιο ή ερώτηση, όπως θέλετε πείτε το. Και αυτό είναι το ότι γίνεται η προσπάθεια να κινηθούμε προς μια πιο πράσινη οικονομία ή όπως θέλετε ας το αποκαλέσουμε. Εσείς πόσο βλέπετε ότι θα πρέπει να τεθεί η έμβαση στους πράσινους δείκτες. Διότι αυτή είναι η βάση, οι πράσινοι δείκτες για το πώς θα μετρήσουμε και θα αξιολογήσουμε αυτό που πρέπει να επιτευχθεί και τους, ε, τις δράσεις και τους στόχους. Τελευταία μου ερώτηση. Οι δείκτες αυτές ε, θα λειτουργούσαν αυτόνομα αντί για στόχους ή μετρήσεις ε, όσον αφορά για παράδειγμα την αξιολόγηση των πόρων για την, τον σχεδιασμό, για παράδειγμα, μιας α, κατεύθυνση ή των δημόσιων προμηθειών. Θα έπρεπε να συζητήσουμε για τα μέσα προς αυτή την πορεία. Ευχαριστώ και αυτή θα ήταν και η δική μου ερώτηση πάνω κάτω. Έχουμε στόχους ε, ε, έχουμε στο Κανκούν καταλήξαμε σε μια συνένεση για δύο βαθμούς αύξηση της θερμοκρασίας και τροχοπέδηση στους δύο και για τους στόχους για το Ρίο που πρέπει να εξειδικεύσουμε περισσότερο αυτή την κατεύθυνση για την αηφορία. Είναι αυτή επαρκής καλή στόχη ή όχι. Δυστυχώς θα πάρουν δύο λεπτά ο καθένας και γι' αυτό πρέπει αντίστροφα να ξεκινήσουμε για να έχουμε δηλαδή αρκετό χρόνο για το επόμενο πάνελ. Παρακαλώ εσείς. Uh, να σχολιάσω το θέμα της πρόθεσης του ρόλου των γυναικών. Πράγματι έχουν ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου ο πρέσβης Βεμέρ αναφέρθηκε σε δύο πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για να διαβριθεί ο ρόλος των γυναικών στην οικονομία και να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση για τις γυναίκες στην έρευνα και την τεχνολογία. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν για την κάλυψη των αναγκών και των γυναικών. Τίθεται βέβαια το θέμα των επενδύσεων. Δεν είναι εδώ το βασικό θέμα συζήτησης, αλλά είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε έτσι ώστε αυτές οι επενδύσεις να στοχεύουν και στις γυναίκες. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν δρόμοι να μπορέσουμε να ωφελήσουμε τις κοινότητες, τις οικογένειες και την κοινωνία στο σύνολό της, στοχεύοντας τις γυναίκες. Οι παράμετρος λοιπόν γυναίκες είναι κομβική παράμετρος. Να τελειώσω λέγοντας ότι στις συζητήσεις άκουσα για κάποιες ε, αναφορές να γίνονται για τη συμμετοχή των γυναικών. Αυτό δεν είναι επαρκές το πράσινο βιβλίο σαν παράδειγμα που δεν είναι τμήμα αυτής της Επιτροπής αλλά συνδέεται με τα θέματά σας είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο προσεκτικότερης εξέτασης στο μέλλον ε, και για την κοινωνική του διάσταση και για τα οικονομικά του ωφέλη. Ευχαριστώ κύριε Ρόχας. Ο Πίτερ. Για τους δείκτες, λέει ο κ. Πίτερ Γούντερς, νομίζω ότι η συνένεση η οποία κρατεί είναι ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα να υπάρξουν κοινοί παγκόσμια δείκτες που θα προσμετρήσουν το λεγόμενο πράσινο ΑΕΠ. Το κοιτάμε αυτό εδώ και χρόνια και δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Θέλουμε συγκεκριμένους μικρότερες εμβέλειας δείκτες σε συγκεκριμένους τομείς. Σαν παράδειγμα στον τομέα της μεταρρύθμισης ε, των επιδοτήσεων συγκρίνουμε τις τιμές που ε, βγαίνουν στους καταναλωτές και μπορούμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο σε διεθνές επίπεδο. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε ένα διατομεακό πράσινο δίκτυ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ανατομέα λοιπόν και αναδράση έχουμε ανάγκη ε, αποτελεσμάτων για τον ρόλο των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να στοχεύσει κανείς το όπου οι κοινότητες ε, ηγούνται της συζήτηση και θεωρούν αυτές τμήμα της λύσης. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα πρέπει όμως να γίνουν. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ασχολήθηκα πάρα πολύ και με την τσιμενοβιομηχανία και με τη χαλιβουργία. Οι πολιτικοί θα πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις βιομηχανίες, να καταλάβουν γιατί οι βιομηχανίες παίρνουν τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν, πού επενδύουν, σε ποιες χώρες και σε ποια είδη τεχνολογιών και εκεί μπορεί να τεθεί το θέμα πλέον σε μια δεύτερη βάση, ε, θέμα κριτηρίων για την πράσινη οικονομία κτλ. Πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί να κατανοήσουν τις ανάγκες των βιομηχανιών, να διαβουλευτούν με αυτές και να ακούσουν τις γνώμες τους. Και για τον ρόλο των γυναικών, συμφωνώ, είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, και εδώ τίθεται το θέμα και στη συζήτηση για τις επιδοτήσεις σχετικά με τον καθορισμό των τιμών της ενέργειας για τις φτωχές κοινότητες, τίθεται το θέμα των γυναικών, τίθεται το θέμα της μεταφοράς αρευστών, τίθεται το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας. Ε, το θέμα όμως δεν είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι η διάρκεια ζωής ορισμένων ε, και το τι συμβαίνει για τη διάρκεια ζωής, κατά τη διάρκεια ζωής ορισμένων προϊόντων όπως ο χάλιβας και το αλουμίνιο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η αναφορά στην αποτελεσματικότητα. Εμείς οι ίδιοι μιλάμε για την αποτελεσματική χρήση των πόρων στα πλαίσια της προσπάθειάς μας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας κατανοούμε επίσης ότι δεν είναι επαρκές να γίνει κανείς πιο αποτελεσματικός, το να παράγει κανείς οθόνες τηλεόρασης πιο αποτελεσματικά, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να γεμίσω με τηλεοράσεις ε, ε, τα δωμάτια του σπιτιού μου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτός, αυτό το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο δεν θα με οδηγήσει πουθενά. Μερικές φορές λοιπόν θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από την απλή έννοια της αποτελεσματικότητας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πράγματι την σπάνη η οποία χαρακτηρίζει ορισμένους πόρους θα πρέπει να δούμε επίσης και ποιος θα είναι ο ρόλος τον οποίο θα πρέπει να κοινοποιήσει πλέον η Ευρώπη προς τα έξω, τον οποίο καλύτερα να παίξει σε σχέση με τέτοια θέματα και θα συζητηθεί ήδη το Σεπτέμβριο ε, ε, φέτος έτσι ώστε να έχουμε πραγματικές συζητήσεις για 20 ε, συν, για το λεγόμενο 20 συν. Χρειάζονται οι δείκτες, συμφωνώ, χρειάζονται οι δείκτες αυτοί τους οποίους έχουμε σχεδιάσει και από οικολογικής πλευράς, περιβαλλοντικής πλευράς, να μιλούν όμως την ίδια γλώσσα με όλους τους άλλους δείκτες. Αν οι περιβαλλοντικοί μας δείκτες δεν είναι εκφράζονται, δεν είναι εκπεφρασμένοι ε, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια σταθμά με τους άλλους δείκτες τότε φοβάμαι ότι δεν θα μας αντιμετωπίσουν σοβαρά. Θα πρέπει να είμαστε στο ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας και θα πρέπει ίσως να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν να ενταχθεί στα λογιστικά μιας επιχείρησης το εξωτερικό κόστος των παραγωγικών του δραστηριοτήτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά την, την σωστή εφαρμογή των βασικών αρχών λειτουργίας. Λοιπόν, καλή Ευχαριστούμε. Καλή τύχη με την πράσινη εβδομάδα και για την νομοθεσία για την, τα λογιστικά για το περιβάλλον του περιβάλλοντος τον Ιούνιο και στο Συμβούλιο θα ξεκινήσουν νέοι τέτοιοι λογαριασμοί λογιστικά να συμπεριλαμβάνουν και τα θέματα του, της συνιστόσα του περιβάλλοντος. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να δώσω συνέχεια να απαντήσω σε δύο σημεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η πράσινη οικονομία και πραγματικά αναζητούμε μεταφορικά να μπορέσουμε να αντανακλάται η συζήτηση με τον σωστότερο τρόπο. Και δεν είναι το θέμα της υποοικονομίας, είναι το θέμα η εναλλακτική οικονομίας. Είναι πώς θα αλλάξει η σημερινή οικονομία ώστε να είναι πιο αηφόρος στο μέλλον. Και ο τρόπος με τον οποίο αρθρώθηκε αυτή η αρχή της πράσινης οικονομίας υπό το πρίσμα της έκθεσης που ο Πίτερ και ε, θεσμικά όργανα και άλλοι συνεισέφεραν. Δεν είναι ένα νιρβάνα, ένας παράδεισος ε, περιβαλλοντικός για αυτόν τον πλανήτη. Είναι η προσπάθεια να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και η διάσκεψη του ρίου είναι μια αναπτυξιακή διάσκεψη, είναι μια διάσκεψη για την ανάπτυξη. Η επικέντρωση όμως είναι πώς θα μπορέσει η πρόκληση της αηφορίας να αντιμετωπιστεί. Αν πάτε στην Παγκόσμια Τράπεζα και ε, παρακολουθήσετε μία ε, συνεδρίαση θα δείτε διαφορετικά θέματα. Εδώ είναι το θέμα στο Ρίο η αηφορία και η δυνατότητα επίτευξης της αηφορίας και αυτό είναι στο επίκεντρο. Ένα από τα πράγματα που θα έλεγα ότι έχουν τεράστια σημασία προσπαθώντας να αρθρώσουμε τους στόχους και την έκβαση που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να διασφαλιστεί ότι χώρες που δεν είναι σε θέση ακόμα να παράσχουν τις ε, βασικές υποδομές για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών τους πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομίες θα δίνουν θέσεις απασχόλησης ε, για τους ε, πολίτες και τα διεθνή συνδικάτα πώς είναι πρωταγωνιστές σε αυτόν τον ρόλο είναι κάτι το οποίο με ικανοποιεί διότι πρέπει να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση και οι επιχειρηματίες και στον ιδιωτικό τομέα και πώς εκείνοι προσπαθούν να δημιουργηθεί μια αγορά στην οποία θα είναι παραγωγή οι ίδιοι για την πράσινη οικονομία και να μην είναι μόνο οι εξορίσσοντες, οι εκμεταλλευτές και δεν έχουμε εδώ τον κρατικό κατά του ιδιωτικού τομέα. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και εδώ θέλω να, πω, να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Ζέμπερ, να επικεντρωθούμε σε μικρή εμβέλεια σε προγράμματα και ε, σχέδια. Αυτό είναι ε, απόλυτα θεμελιώδη περίοδες ε, για τη μετάβαση. Οι μεταβατικές, οι μεταβάσεις και αλλαγές που βλέπουμε σύμφωνα σήμερα και η μετακίνηση προς μια μεγαλύτερη ε, οικονομία της γνώσης. Πρέπει να δούμε την συνολικότερη εικόνα. Αν θέλουμε οι αναδυόμενες, αναπτυσσόμενες οικονομίες να επενδύσουν σε μια διαφορετική οικονομία στο μέλλον, δεν έχουμε μόνο τα προγράμματα grassroots ε, για τους ίδιους τους πολίτες. Θα δούμε ένα παράδειγμα, την Κένια. 80% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε εξηλεκτρισμό ε, έχει περάσει το θέμα της ε, ε, και θα περάσει σε τριπλασιασμό των υποδομών χωρίς να εκλείεται ούτε ένα γραμμάριο άνθρακα εντό εισαγωγικών με αιωλική και πράσινη ενέργεια. Για να επιτευχθεί αυτό θα χρειαστεί υποστήριξη για τις υποδομές και την πρόσβαση στις οικονομικές δυνατότητες. Είναι όμως ικανή να τα καταφέρει η Κένια και βλέπουμε εδώ μια χώρα και αυτό είναι ε, η, η λογική πίσω από την συνεργασία και την ανάπτυξη. Ένα δις ε, Αφρικανών ή θα ακολουθήσουν την πορεία των τελευταίων δεκαετιών και τότε δεν θα υπάρχει ευκαιρία να επιτευχθούν οι στόχοι για το περιβάλλον που θέλουμε να επιτύχουμε ή θα πρέπει να μετακινηθεί σε νέες υποδομές προς μια νέα κατεύθυνση η Αφρική στον 21ο αιώνα. Είναι η μόνη ευκαιρία που έχει και έτσι κλείνει ο κύκλος για την ανάπτυξη, για την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και να μην το ξεχνάμε αυτό στο Ρίο, επιτέλους για μια φορά ας αρχίσουμε να προσπαθούμε να μην κατηχούμε ο ένας τον άλλον τι πρέπει να κάνουμε στις χώρες μας. Ας επανέλθουμε στην αρχική ιδέα της διεθνούς συνεργασίας. Είσαστε εσείς μια κυρίαρχη χώρα. Εγώ έχω συμφέρον να αναπτυχθείτε. Ας δούμε από κοινού πώς μπορούμε να συνεργαστούμε να, θα, δεν θα πρέπει να λέμε στους άλλους ή να προσπαθούμε να τους επιβάλλουμε το τι πρέπει να κάνουν. Θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας υπό το πρίσμα μας. Να βοηθηθεί η διεθνή κοινότητα να κινηθεί προς αυτούς τους στόχους για την επίτευξη της ε, παγκόσμιας αηφορίας και ανάπτυξης και για την επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη και το πάνελ, το φόρουμ για την αηφορία, εξετάζοντας αν είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Αυτός θα ήταν ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση. Για τις γυναίκες εν τέλει θα ήθελα να πω δύο λόγια. Εσείς οι γυναίκες και τα Ηνωμένα Έθνη και από πλευρά των θεσμών προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθείτε στο Ρίο, να διασφαλίσουμε ότι η προοπτική της αηφορίας στην ανάπτυξη με ηγέτιδες γυναίκες και τη συμμετοχή τους ε, δεν θα ε, διεξαχθεί μόνο μια περιθωριακή συζήτηση επ' αυτού αλλά θα βρεθούν στο επίκεντρο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι, ευχαριστώ. Θα είναι πραγματικά συναρπαστικό το εγχείρημα σε παγκόσμιο επίδημα να προσπαθούμε να βρούμε δείκτες για την ευημερία και την ανάπτυξη προς αυτή την πορεία. <clears throat> Πέρα από το παραδοσιακό ΑΕΠ ως ε, γνώμονα ως πύχη. Η αηφορία ας πούμε είναι η κύρια έννοια υπό την οποία πρέπει να κινητοποιηθούμε, αλλά να είμαστε πιο εξειδικευμένοι σε σχέση με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και τους δείκτες που θα μας βοηθήσουν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που πρέπει. Εξαιρετική ήταν αυτή η δουλειά του πρώτου γύρου, του πρώτου πάνελ. Σας ευχαριστώ για το ότι συνεισφέρατε στο να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Θα επανέλθουμε και θα ξανασυναντηθούμε υπό τη μία ή άλλη σύνθεση και στο ένα ή άλλο όργανο πριν από το Ρίο ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσκαλώ τώρα τους συμμετέχοντες στο δεύτερο πάνελ να έρθουν στο Προεδρείο και θα συνεχίσουμε άρρηκτα τη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εν τω μεταξύ Θα ήθελα να κάνουμε κάτι, να πω στα μέλη να περάσουν να δουν το πρώτο ηλιακό αεροπλάνο, το μόνο το οποίο υπάρχει σήμερα παγκόσμια που ήρθε από την, από την ε, Ελβετία στις Βρυξέλλες και μετά από αυτή τη συνεδρία στις 12.30 θα περιμένει ένα πούλμαν στη Ντάρνεμ, που θα είναι μπροστά στο Άτριουμ και που θα, θα μας οδηγήσει, θα μας πάει στο ηλιακό αυτό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο. Ενδιαφέρον θα είναι για πολλούς από εμάς να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με εκείνους που δημιούργησαν με ιδιωτικά κονδύλια ένα ηλιακό αεροπλάνο που κινείται με την ε, ε, ηλιακή αυτή ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συναποτελούντες στο δεύτερο πάνελ αφήχθησαν και μπορούμε αμέσως να συνεχίσουμε τις εργασίες μας με την συζήτηση για την αηφορία στην ανάπτυξη και την διακυβέρνηση της αηφορίας στην ανάπτυξη. Πώς μπορούμε από πλευράς διαρθρώσεων και θεσμικών οργάνων να τα πετύχουμε όλα αυτά. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω και πάλι τον Μπρίς Λαλόντ. Τώρα είσαστε ο εκτελεστικός συντονιστής για το Ρίο Γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια στο κίνημα υπέρ του περιβάλλοντος και τα Υπουργεία για το περιβάλλον. Υπουργεία Περιβάλλοντος είναι ένα σε εξέλιξη με μεταξελισσόμενο διακόσια σε θέμα. Παρακαλώ έχετε τον λόγο για να κάνετε την εισαγωγή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Όπω γνωρίζετε το ορίο ΣΥΝ 20 βασίζεται κυρίω στι ε, πρωτοβουλίες των χωρών. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συζήτηση. Ε, περιμένουμε όμω ακόμα περισσότερες ε, ε, πληροφορίες και απόψεις από ό,τι έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. <clears throat> Ίσως να πρόκειται για έλλειμμα ηγεσία και χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω από αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ιστορικό ε, ανάληψη ηγετικού ρόλου σε τέτοιες καταστάσεις. Εσείς είστε μέλη των επιτροπών, των πολιτικών ομάδων και ε, περιμένουμε περισσότερα από εσάς. Ε, κύριο χαρακτηριστικό των ε, προσπαθειών μας είναι ότι εστιάζουμε κυρίως ε, στα βραχυπρόθεσμα μέτρα και όχι τόσο στα μακροπρόθεσμα, γιατί δεν έχουμε την ολιστική προσέγγιση που αρμόζει. Μάλλον και γιατί εστιάζουμε τόσο πολύ στην παρακολούθηση, επιτήρηση δημοσιονομικών κτλ. Ε, στην ε, διεθνή διακυβέρνηση λοιπόν, αν ήμασταν ακριβείς, θα έπρεπε να συνδυάσουμε το, το G20 με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Στην βιωσίμη ανάπτυξη, με κυρίως την ανάπτυξη. Πρώτα πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε την, τις επιτυχίες της ανάπτυξης. Πολλές, πολλοί θεσμοί και οργανισμοί υπάρχουν για την ανάπτυξη, αλλά είναι αποδοτικοί, είναι ακριβείς εστιάζουν στο, τι παράγει μια χώρα, στο τι κάνει μια χώρα και στην διάδραση με την παγκόσμια οικονομία. Η Επιτροπή θα έχει μια ανακοίνωση ε, από κοινού από, το, από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ε, και Οικονομίας. Και το χρειαζόμαστε αυτό. Είναι απαραίτητο γιατί υπάρχουν αυτά τα σταγανά μέχρι τώρα ανάμεσα στους δύο τομείς. Ε, από την άλλη, ε, ο τομέας της ε, ενέργειας και του περιβάλλοντος όλα είναι και περισσότερο ασχολείται με την ανάπτυξη. Αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν, στήριξη στην ανάπτυξη. Εκατό δις ε, το χρόνο από το 2020 λέμε. Εντάξει, αλλά πώς θα τα βρούμε αυτά. Πώς θα έχουμε έτσι, την καινοτομία στη χρηματοδότηση. Αυτό είναι κέρια σημασία ζήτημα και μάλλον γύρω από αυτό θα στραφεί και η συζήτηση. Δεύτερον, αηφορία, η βιωσιμότητα. Ξέρετε το δίκτυο δημιουργήθηκε στη Στοκχόλμη το 1982, αλλά πιο πριν και το 87 είχαμε αντίστοιχε ε, διαδικασίες και το 92 ε, με ενδιαφέρουσε συγκυρίε μετά την πτώση του ε, του Βερολίνου. Και το Ρίο δημιούργησε το CSD, Επιτροπή βιώσιμη Ανάπτυξης. Ε, βέβαια τώρα σε διεθνή φόρουμ δεν μπορούμε να αναφερόμαστε πλέον μόνο σε ανάπτυξη, αυτό ήταν ο όρο δημιουργίας του CSD. Ε, προσπαθεί να ε, συγκεντρώσει διαφόρους, ε, διαφόρα ενδιαφερόμενα μέρη και έχουμε πλέον εννέα κύριες ομάδες. Μιλήσαμε για, το, την, για την διάσταση του φύλου, αλλά για παράδειγμα δεν μπορούμε να έχουμε διακυβέρνηση και πράσινη οικονομία χωρίς τοπική διακυβέρνηση και την επιχείρηση χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή ε, των ε, κυβερνητικών αποφάσεων και δεν έχουμε καταφέρει να τους συμπεριλάβουμε όλους αυτούς τους φορείς ε, στην διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η βιώσιμη ανάπτυξη όμως αφορά και κάτι όπως την διάσκεψη όρους που για παράδειγμα έχει υπογραφεί μόνο από 30 φορείς. Βέβαια αφορά μόνο ε, κράτη. Αλλά εδώ και πολύ καιρό είχαμε πολλές πρωτοβουλίες και εκθέσεις από επιχειρήσεις. Τι κάνουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, πού πάνε, ποιος τις αξιολογεί. Αυτά χρειαζόμαστε, ούτω ώστε αυτές οι εκθέσεις να έχουν κάποιο σκοπό. Ε, υπήρχε και ένα δόγμα στις, στα Έθνη ανάμεσα στις λειτουργικές ε, οντότητες και στις ε, απλές ε, οντότητες. Ε, πολλοί λένε ότι δεν μπορούμε πλέον να, ε, κάνουμε να αγγίξουμε την ε, χάρτα γιατί έτσι θα ανοίξουμε ε, το κουτί της Παντόρας. Αλλά όλα αυτά τα θεσμικά ζητήματα συνδέονται και με τις ιδέες μας για το πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Οι Βραζιλιάνοι θέλουν να δημιουργήσουν μια οργάνωση ομπρέλα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός ήταν στόχος του CSD. Όμως, τι πήγε στραβά. Όταν ξεκίνησε ήταν όλα τέλεια και ρόδινα. Τώρα όμως λένε ότι ε, έχει γίνει υπερβολικά, στρέφεται υπερβολικά στα τεχνικά ζητήματα. Βέβαια, όπως ξέρετε, δεν είναι δεσμευτικό. Τίποτα δεν είναι δεσμευτικό. Ε, για να υπάρχει κάτι δεσμευτικό πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση. Και το θέμα είναι, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι βάση συμφωνίας γιατί ξέρετε ότι μετά το ε, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλοι θεωρούσαν ότι ο προστατευτισμός ε, ήταν κάτι πολύ κακό, ενώ το, το εμπόριο ήταν αυτό στο οποίο θα πρέπει να βασίσουμε τις οικονομίες μας. Βέβαια, βλέπετε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή, θα μας πάρει πολλούς ε, γύρους όλοι αυτοί ο γύρο ειδίκησαν στη λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Α κάνουμε το ίδιο λοιπόν. Α έχουμε γενικέ συμφωνίε στη βάση με ανάπτυξη, στην, ε, στο περιβάλλον και τη βάση στην οικονομία. Ε, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα λοιπόν και εδώ. Θα έχουμε γύρου, ε, διαφόρου, ε, μία για τα λογιστικά ζητήματα, μία το περιβάλλον δηλαδή πώς να έχουμε ε, πράσινα στοιχεία στο ΑΕΠ. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να γίνουν λοιπόν. Ένας γύρος για την ενέργεια. Ξέρουμε τι να κάνουμε, έχουμε την έκθεση Γιάνν Κέλλερ. Τα έχουμε όλα αυτά επιτάπητος, μπορούμε να θέσουμε στόχους. Μετά έχουμε τη γεωργία. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να έχουμε κάτι πιο ισχυρό, μια συμφωνία ε, με, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δεσμευτούν τα κράτη. Το Ρίο δεν θα επιλύσει τα προβλήματα του κόσμου, θα θέσει όμως α στρώσει το δρόμο ε, για τα επόμενα 20 χρόνια. Το έργο, στο πλαίσιο ε, των ΟΕΕ είναι κατακαιρματισμένο γιατί δεν υπάρχει ε, καθολική ιδιότητα μέλους στη UNEP. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα με το UNEP, οι υποχρεωτικές ε, συνεισφορές, γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτική συνεισφορά, γίνεται εθελοντικά. Άλλο πρόβλημα είναι η σύνδεση με τις συμβάσεις. Οι συμβάσει αυτέ βρίσκονται σε ένα ξεχωριστό μονοπάτι. Πώ μπορεί να υπάρχει συντονισμό. Γιατί ε, δυσκολεύονται πολύ αναπτυσσόμενε χώρε ε, για να καλύψουν αυτέ τι ε, δεσμεύσει και τι προποθέσει. Ένα διπλωμάτη από αναπτυσσόμενε χώρε πρέπει να ταξιδέψει 10 φορέ παραπάνω από του υπόλοιπου. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε αυτό το σύστημα πιο αποδοτικό. Ε, ήταν ένα όρο που άκουσα προηγουμένω. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν μια, έναν οργανισμό ε, με δύο ε, φόρα, ένα για τα κράτη-μέλη και ένα για τις επιτροπές αυτές. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θέλει η UNEP να ε, μετατραπεί σε έναν οργανισμό. Αυτό βρίσκεται σε στάδιο συζητήσεων. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη διεξάγουν μία μελέτη γιατί λένε ορισμένοι ότι αν αυξήσουμε τον περιβαλλοντικό πυλώνα τότε τι γίνεται με τον κοινωνικό πυλώνα. Αλλά αυτό σχετίζεται και με τον ILO. Τι θα γίνει λοιπόν αυτό το θέμα δεν μπορούμε να έχουμε πράσινη οικονομία χωρίς να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Στη διακυβέρνηση βέβαια έχουμε ε, δίκαια, πρότυπα και ούτε καθεξής. Είναι σημαντικό η, Ευρώπη, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 να επιφέρει αλλαγές στην ε, καθημερινή ζωή ε, του κόσμου. Το Ρίο θα μιλήσουμε για τους ωκεανούς. Πολύ σημαντική για πολλά νησιά. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την πράσινη οικονομία, λένε κάποιοι, αλλά και για την ε, γαλάζια οικονομία, την μπλε οικονομία. Και αυτό γύρει το ζήτημα της διακυβέρνησης. Δεν θα αναφερθώ τώρα στις αρχές του Ρίου, αλλά υπάρχει μία αρχή. Η μη... Μη οπισθοδρόμηση. Θα πρέπει λοιπόν να γινόμαστε καλύτεροι και καλύτεροι. Ε, υπάρχει όμως ο κίνδυνος αυτή τη ε, ε, όταν προστατεύουμε το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπρίσλα Λάντ, για αυτή την εισαγωγή σε αυτού του γύρου, σε αυτό το πάνελ, με πολύ μεγάλο εύρος προβληματισμού και σκέψεων για τις δομές, για την παγκόσμια διακυβέρνηση, για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε όλα αυτά και τι θα σημαίνει αυτό όταν θα βελτιωθεί η UNEP και τι θα συνεπάγεται αυτό για τα άλλα θεσμικά όργανα και τις περαιτέρω βελτιώσεις. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από την Καλαβρία, από τον συνάδελφό μας ε, Πυρίλο έχουν προσκληθεί. Καλώς ήρθατε, ευπρόσδεκτοι είσαστε να παρακολουθήσετε αυτή τη συζήτηση. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε στο πάνελ. Καλωσορίζω και πάλι τώρα τον Ρικάρδο Νέιβα Ταβάρες, πρέσβη της Βραζιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς είσαστε οι αμφιτρίονες αυτής της πρώτης διάσκεψης κορυφής, συνόδου κορυφής και φυσικά η αμφιτρίων χώρα είναι πραγματικά ιδιαίτερα φιλόδοξη. Ακούσαμε από τον Μπρίσλα Λάντ σε σχέση με μια οργάνωση, ε, ένα οργανωτικό πλαίσιο εγίδας ή ομπρέλας ε, φιλόδοξο για την προώθηση αυτών των στόχων υπό την δική σας ακριβώς ε, υποδοχή. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμη ε, κύριοι συμμετέχοντε ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντο Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτών για την πρόσκληση αυτή να έρθω και να συζητήσω τι κύριε γραμμέ τη διάσκεψη των εθνών για την αηφορία στην ανάπτυξη που θα γίνει τον Ιούνιο 2011 στο Ρίο Ντεζανέιρο. Όπω μπορείτε να φανταστείτε είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη Βραζιλία. Όχι μόνο επειδή εμεί θα είμαστε οι αμφιτρίωνε αυτή τη διάσκεψη 20 χρόνια μετά τη διάσκεψη των ΗΕ για το περιβάλλον και την ε, ανάπτυξη πάλι στο Ρίο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι παραδόσεις τη Βραζιλία και τι δεσμεύσει τη διεθνείς προσπάθειες να εκφραστεί με συγκεκριμένο τρόπο ο στόχος και τα μέσα τη αηφορία στην ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερη ικανοποίηση για μένα να μπορώ να σα προσφωνήσω για αυτό το θέμα όπως έχω κάνει ήδη στο παρελθόν με άλλε αφορμές στην ΕΚΟΣΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, ε, όπως ίσως θα θυμόσαστε. Τότε ε, το ψήφισμα 64 236 ήταν ένα σχέδιο για ε, υποσυζήτηση σε σχέση με την Νέα Υόρκη και που είχε ξεκινήσει η ιδέα του να αναλυθεί η διάσκεψη Ρίο 20 με την έναρξη της ε, Γενικής Συνέλευσης ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, τότε το 2007 συνεργαστήκαμε πάρα πολύ εκ του και όλοι γνωρίζουν ότι το ψήφισμα 64 236 ενσωμάτωνε τα μελήματα της ανησυχίας της Ευρώπης για την αηφορία στην ανάπτυξη και τους κυριότερους στόχους για, για, αυτό, για αυτή την προσπάθεια. Αυτά που συζητάμε σήμερα. Πράσινη οικονομία στην αηφορία της ανάπτυξης, εκρίζωση της φτώχειας, θεσμικό πλαίσιο για την αηφορία στην ανάπτυξη. Πρωτού εν, επικεντρωθώ στα κυριότερα θέματα, επιτρέψτε μου να πω μόνο δύο λόγια για τις προσδοκίες μας πριν από αυτή τη διάσκεψη. Όταν υιοθετήθηκε αυτό το ψήφισμα, η Γενική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε ότι η διάσκεψη θα στόχευε στο να ανανεώσει την πολιτική δέσμευση υπέρ της αηφορίας στην ανάπτυξη. Θα αξιολογούσε τις προόδους και τα κενά στην υλοποίηση των προηγουμένων προσπαθειών και θα εντόπιζε νέα αναδιόμενα θέματα. Τώρα, για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων Ήδη το 1992 όταν τότε υιοθετήσαμε τα κυριότερα μέσα με τη διακήρυξη του Ρίο την ε, ημερήσια διάταξη του 21ου αιώνα, τις κλιματικές αλλαγές και τη σύμβαση για τα ε, θέματα της ε, ε, καταπολέμησης της απερίμωσης. Το Ρίο Συνήκωση πρέπει να βασίζεται σε αυτά τα ισχυρά θεμέλια, καθώς επίσης ε, και σε μια πλήρη ημερήσια διάταξη για την επίτευξη των στόχων, για να δημιουργηθεί μια ημερήσια διάταξη για το μέλλον, για την εφορία στην ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα ελπίζουμε ότι το έγγραφο το οποίο ε, οι αποφάσεις που θα υιοθετηθούν θα εγκριθούν ε, στο Ρίο πράγμα που είναι υποδιαπραγμάτευση από το Προεδρείο και τους συμμετέχοντες, θα δίνουν πολιτικές κατευθύνσεις που θα είναι αξιόπιστες και πραγματικά να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν. Η συζήτηση σε θεσμική βάση της διακυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεσα πρακτικά αποτελέσματα, όπως την αναθεώρηση της εφαρμογής των ε, διεθνών συμβατικών δεσμεύσεων. Στρέφομαι τώρα στο κύριο θέμα που είναι υποσυζήτηση. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η κύρια πρόκληση που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την αηφορία στην ανάπτυξη είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε και να πετύχουμε τι λύσει για τα προβλήματα συνεκτικότητας και συνοχής και συντονισμού και για την καλύτερη λειτουργία των ε, θεσμικών οργάνων και των ε, μέσων και εργαλείων που εμπλέκονται στην ε, αηφορία στην ανάπτυξη, όπω το πρόγραμμα των ΗΕ για την Ανάπτυξη, καθώ επίση και την Επιτροπή για την Αηφορία στην Ανάπτυξη, το Συμβούλιο για την ανάπτυξη, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνή Οργανισμό ε, Εργασίας, ε, καθώς επίσης ε, και πολλά άλλα θεσμικά φόρα. Για να διευρυνθεί λοιπόν θεσμικά η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αξιολογήσουμε και την εντολή και τις επιδόσεις των υφισταμένων θεσμικών οργάνων. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε χρόνια προβλήματα των σημερινών θεσμικών συσχετισμών όπως την έλλειψη η στενότητα κεφαλαίων και να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο τι απαιτήσει ε, που τίθενται ενώπιόν μα για την επίτευξη τη αηφορίας στην ανάπτυξη. Μετά την 1η Νοεμβρίου, που είναι η προθεσμία από απο πλευρα ε, των προτάσεων εθνικών ε, εισφορών, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουμε καλύτερα τι εναλλακτικέ λύσει για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την αηφορία στην ανάπτυξη. Ήδη γνωρίζουμε κάποιε από τι προτάσει και τοποθετήσει των διαφορετικών εμπλεκόμενων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει δημιουργία ενός περιβαλλοντικού οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που θα χρησιμοποιεί ακριβώς ε, ε, τους οργανισμούς, τα θεσμικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη σε σχέση με την εμπλοκή και δέσμευση αύξησης κονδυλίων, παρότι δεν έχουμε κάποια αντίρρηση σε σχέση με την αλλαγή εντολής, είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τα κονδύλια. Χώρες όπως ε, η Ελβετία και άλλες ε, και διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι υπέρ του να υπάρξει ένας παγκόσμιος μηχανισμός για την αναθεώρηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που θα είναι παράλληλη με την εντολή όσον αφορά την λειτουργία του Συμβουλίου. Η ε, συνδιάσκεψη για την ανάπτυξη των ΗΕ πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί αυτό το παγκόσμιο επίπεδο σε συνδυασμό με το περιφερειακό και τοπικό ώστε να ενδυναμωθούν οι μηχανισμοί σε όλα τα επίπεδα. Οι προτεραιότητε θα πρέπει να καθορίζονται εκ των κάτω προ τα άνω και αρρωγή θα πρέπει να προσφέρεται ώστε να προχωρήσουμε. Η βραζιλιανική κυβέρνηση έχει και εκείνη κάποιες συγκεκριμένε ιδέες ε, επ' αυτών των θεμάτων. Όπως ε, θα έχετε συνειδητοποιήσει, έχουμε και το θέμα της δημιουργίας ε, μιας δυνατότητας ε, στέγασης υπό συγκεκριμένη αιγίδα ή ομπρέλα αυτών των δράσεων. Ποιοι είναι οι λόγοι για αυτές τις προτάσεις μας. Πρώτον, θεωρούμε ότι αν επιθυμούμε καλύτερη διακυβέρνηση σε παγκόσμιο πλαίσιο για την εφορία της ανάπτυξης πρέπει να ενδυναμωθούν οι κανόνες του, της ε, ΕΚΟΣΟΚ, ενός από, τους, ε, ένα, ενός από τα κύρια σώματα. Πρέπει ο περιβαλλοντικός τομέας να μπορέσει να ενδυναμωθεί. Αυτό το πρότυπο θα διασφαλίζει όσον αφορά τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών στην λήψη απόφαση. Αυτό θα απαιτεί μια τροποποίηση του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή, έναυσμα, ώστε να υπάρξει μια ολόκληρη σειρά αλλαγών και προσαρμογών. Για να δημιουργηθεί αυτό ο πυλώνας των Ηνωμένων Εθνών και να ε, επιτευχθεί η λειτουργία του. Δεύτερον, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα περιβαλλοντικά θέματα δεν καλύπτονται αποκλειστικά από την UNEP και άλλοι φορείς ε, όπως ε, ο Οργανισμός ε, Τροφίμων και Γεωργίας, ε, όπως η UNESCO, έχουν και οι άλλοι αυτοί οι φορείς σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στο τομέα τους. Η υψηλή ομάδα αξιωματούχων της ECOTOC τα διάφορα φόρα όσον αφορά την διεθνή αυτή προσπάθεια καταδεικνύουν πως η αηφορία στην ανάπτυξη είναι ένα εγκάσιο, οριζόντιο θέμα. Αν αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία εντάξει και τον πυλώνα της αηφορίας, αυτό θα συνεισέφερε στη διαδικασία αναθεώρησης του Διεθνούς Πλαισίου Συνεργασίας, Συνεργασίας για την Ανάπτυξη, λαμβάνοντα υπόψη τις τρέχουσες προτεραιότητε για τα θέματα αυτά. Τρίτον, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η θέσπιση, η συγκρότηση αυτού του μηχανισμού θα μπορούσε να ε, συνεπάγεται πρόσθετα κόστη για τη χρηματοδότηση αυτού του οργανισμού. Υπό έναν οργανισμό αιγίδας ε, συστέγασης θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την λειτουργία αυτή και να διασφαλίσουμε την ε, διαφάνεια και την λειτουργικότητα γραμματείας ε, και λειτουργία των προγραμμάτων. Στεναρά πιστεύουμε όπως και πολλές άλλες χώρες ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει την ενιολογική αυτή προσέγγιση και προσπάθεια υπερβελτιώσεων ώστε να επιτεθούν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα προηγούμενα 20 χρόνια. Δεν θα θέλαμε σε σχέση με την ε, αηφορία να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με διαφορετικούς πυλώνες ε, σε σχέση δηλαδή με τον οικονομικό, ε, κοινωνικό, περιβαλλοντικό τομέα. Και δεν θα έπρεπε να έχουμε κατακαιρματισμό ή οπισθοδρόμηση, τομεακά μόνο αντιμετωπίζοντας θέματα περιβάλλοντος ή αηφορίας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε και να εξετάσουμε αυτή την ιδέα μια συστέγαση κοινή αιγίδα ή ομπρέλα σε ένα διεθνέ πλαίσιο για την αηφορία στην ανάπτυξη με ελαστικότητα. Ουσιαστικά θα θέλαμε να επιτρέψουμε μια επίσημη πρόταση να εντάσει την μετεξέλιξη των συζητήσεων επιτόπου ώστε να ευδοκιμήσουν. Όπω γνωρίζετε, ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών το 2010 δημιούργησε μια ομάδα υψηλών αξιωματούχων για τα θέματα αυτά. 20 προσωπικότητες τη συναπατίζουν, όπως ο πρώην η, κυρία Γκρο Μπρούντλαντ, πρώην Πρωθυπουργό τη ε, Νορβηγία ε, και άλλοι. Το έργο αυτού του πάνελ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο τη, ε, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2011. Και έτσι θα μπορούσαν να υπάρχουν, να υπάρχουν αξιόλογε συνεισφορέ σε σχέση με τα θέματα υποδιαπραγμάτευση στο Ρίο. Θα θέλαμε επίση να υπάρξει μια αυξημένη συμμετοχή μη κυβερνητικών εμπλεκομένων και φορέων σε αυτή τη συζήτηση γυναικών, νέων, επιχειρηματικών τομέων, κοινωνικών τομέων, με όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμφέρον να εμπλακούν και να συνεισφέρουν σε διεθνές και ε, περιφερειακό επίπεδο. Εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών που είναι θεμελιώδες στοιχείο για τη νέα αυτή κατεύθυνση και την ε, ευδοκίμηση των στόχων. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας και τονίζοντας ότι η Ρίο συν είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναζωογονήσουμε το κληροδότημα, την κληρονομιά του Ρίο στο παρελθόν. Ιδιαίτερα προς επίτευξη κοινή συνένεσης για να προχωρήσουμε σε μια ισόρροπη, ισορροπημένη, ε, συντονισμένη δράση υπέρ του περιβάλλοντος, ε, υπέρ της ε, κοινωνίας και οικονομίας των τριών αυτών πυλώνων για την αηφορία στην ανάπτυξη. Σημαντικό θα είναι σε υψηλότατο επίπεδο στην εκπροσώπηση αυτή στο Ρίο να διασφαλίσουμε διασφαλίσουμε την μέγιστη αποτελεσματικότητα προς όφελος όλων. Ευχαριστώ. Yeah. Um, Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Κύριε Πρέσβη Ταβάρες. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εισήγησή σας. Είναι η τέλεια χώρα η Βραζιλία για να διεξαχθεί αυτή η διάσκεψη και με κάθε σθένος καταβάλλεται προσπάθειες να στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημα. Αναφερθήκατε στην κοινωνία των πολιτών που θέλουμε να εμπλακεί, ώστε οι πολίτες ε, με τον ρόλο που θα αναπτύξουν ε, εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών να εμπλακούν πλήρως. Είναι η στιγμή να καλωσορίσουμε τον Ντέρεκ Όσμπον από πλευρά τη ΕΚΟΣΟΚ υπό αυτή την εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών έχετε ήδη κάνει σημαντικό έργο επ' αυτών. Δώστε μας κάποιες ιδέες ε, για το έργο σας. Έχετε τον λόγο λοιπόν από πλευράς της ε, ΕΚΟΣΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύριε Όσμπο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι καλό όταν η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και να στηρίξει τις εργασίες του Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά. Νομίζω ότι συμβολικά το Κοινοβούλιο πρέπει να διευκολύνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Να ξεκινήσω με αυτά στα οποία αναφερθήκατε σχετικά με το πώς δακτυλοδειχτούμε ή μεν τους δε. Αυτό ίσως δεν είναι πολύ θετικό, αλλά θα πρέπει ίσως να στρέψουμε το δάκτυλο προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Εμείς κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται εμείς να πεσβεύουμε στους άλλους το τι θα πρέπει να κάνουν, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε με το παράδειγμά μας να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σαν τμήμα της προετοιμασίας μας για το θέμα της διακυβέρνησης. Έχει σημασία να προχωρήσουμε, γιατί αν και αυτές οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν κάποια σημασία, το κεντρικό σημείο στο οποίο θα επιδιώξουμε την αηφορία είναι σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, κυβερνήσεων κρατών μελών, που είναι κυρίαρχες σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. και που αν δεν τα καταφέρουν σε εθνικό επίπεδο δεν πρόκειται να τα καταφέρουν και σε επίπεδο διεθνών συμφωνιών. Ε, και βρίσκουμε τέτοια παραδείγματα έλλειψης συνοχής και σε όλες τις χώρες μας. Οι εθνικοί μηχανισμοί για την προώθηση της αηφορίας θα πρέπει να ενισχυθούν εκ νέου. Ένα από τα βασικά θέματα το οποίο έχουμε αναφέρει επανειλημμένα σχετικά με την αηφόρο ανάπτυξη είναι ότι η ατζέντα για την ανάπτυξη αυτή δεν ανήκει μόνο στους περιβαλλοντιστές και τους υπουργούς περιβάλλοντων, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις σε αυστηρά οικονομικό επίπεδο. Οι υπουργοί λοιπόν οικονομικών του κόσμου θα πρέπει να πάρουν μαθήματα στον τομέα αυτό. Μιλάμε για τροποποιήσεις της δομής των συστημάτων φορολογίας, ε, η διαδικασία έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ, με οδυνηρά αργό τρόπο μέχρι τώρα. Πρέπει να πείσουμε τους Υπουργούς Οικονομικών να φύγουν από το συντηρητικό καβούκι τους, κάποιος τους ονόμασε αγιατολάδες της λογιστικής προηγουμένως, και να λάβουν υπόψη τους τα συμφέροντα του λαού τους για την αηφόρο ανάπτυξη. Απαιτείται λοιπόν μεγαλύτερη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο πάντα απαιτούνται και καλύτερες στρατηγικές. Υποτίθεται ότι αυτό βγήκε από το ΡΙΟ. Όλες οι χώρες του κόσμου ανέλαβαν την υποχρέωση να προσπαθήσουν να επιβάλλουν τους νόμους αυτούς, τις αποφάσεις τους μάλλον σε επίπεδο κράτους. Αλλά πάρα πολλές από τις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης είτε απέτυχαν είτε έχουν αρχίσει και σβήνουν σιγά σιγά. Και στο εσωτερικό της Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αηφορία είναι ένα βήμα πριν από το θάνατο. Έχουμε περάσει έτσι και αλλιώς την ξεχάσαμε. Μιλάμε για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων για τη στρατηγική του 2020. Σημαντικό αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα και θα πρέπει να την αναβιώσουμε και να την αναζωογονήσουμε με νέους στόχους. απαιτείται να προσπαθήσουμε να δούμε με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο που παίζουν διάφορα σώματα έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι εμπλεκόμενοι ε, να ακουστούν είτε συμβουλευτικά σώματα είτε συμβούλια συμβουλευτικά τα οποία έχουν αρχίσει να σβήνουν τον τελευταίο καιρό και να μειώνεται η σημασία τους. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν επίσης πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν σε σχέση με την αηφορία. κ. Βάτεμπεργκ και Φάλκεμπεργκ, συγγνώμη, αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να πιέσουμε τις τοπικές αρχές να κάνουν περισσότερα. Ε, μερικές φορές οι τοπικές αρχές κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Είναι ηγέτιδες στον τομέα αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να ακούσουμε τις ιδέες τους και να μπορέσουμε να ε, ε, κυκλοφορήσουμε τα μηνύματά τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο και από αυτούς μπορούν να πάρουν μαθήματα μερικές φορές οι εθνικές κυβερνήσεις έτσι ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για την προσπάθεια προώθησης της αηφορίας. Και εδώ είναι ένα άλλο σημείο της συζήτησης για, <clears throat> το, για τις κυβερνήσεις. Το θέμα του επιχειρηματικού κόσμου φυσικά έχει ένα κρίσιμο ρόλο για να πάνε καλά τα πράγματα, στην προσπάθεια να πάνε καλά τα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες όπως υπόθηκε σήμερα το πρωί. Αλλά νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με τον στόχο τον οποίο πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν την εταιρική, ε, θα έλεγα, την εταιρική αηφορία και σε επίπεδο εσωτερικό και σε επίπεδο συνεργασιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Για το διεθνές επίπεδο, το παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα επαναλάβω σε αυτά τα οποία τίποτα, μετά από αυτά τα οποία ακούστηκαν και από τις οργανώσεις των πολιτών με τις οποίες συνεργάζουμε, θα υποστηρίξουμε όλες τις θετικές ιδέες οι οποίες θα προέλθουν για την ενίσχυση των συμβάσεων αυτών διεθνώς. Το USCND, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη, εν έχει ε, προχωρήσει, έχει κάνει πολλά πράγματα εδώ και 19 χρόνια από την πρώτη συνάντηση στο Ρίο. Και καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε γιατί δεν αποδίδει τόσο σήμερα όσο απέδιδε παλαιότερα. Θα δούμε ότι βασικό είναι οι νέες δομές για την προώθηση της αηφορίας θα πρέπει να εμπλέκουν και τους Υπουργούς Οικονομικών και τους Υπουργούς Εμπορίας εμπορίου, συγγνώμη, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους τα βασικά μέσα για την προώθηση των στόχων μας. Ανεξάρτητα από τις δομές τις οποίες θα δημιουργήσουμε διεθνώς, το θέμα δεν είναι ποιος θα συμμετέχει απλά, αλλά θα πρέπει αυτός που θα συμμετέχει να αντιπροσωπεύει πραγματικά αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν πραγματικές αποφάσεις στον τομέα της φορολογίας, στον τομέα των ε, διεθνών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να ενισχύσουμε και τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και να προσπαθήσουν να συντονιστούν οι υπηρεσίες με καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει επίσης και τις διμερείς συμφωνίες να προσπαθήσουμε να δούμε πώς οι συζητήσεις αυτές πρέπει να ενισχυθούν στο μέλλον δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια επιτροπή που να αντιπροσωπεύει όλα τα σώματα των Ηνωμένων Εθνών και όλους τους θεσμούς των Bretton Woods, του Bretton Woods. Έτσι ώστε να συμπληρώνουν με τη δράση τους ό,τι γίνεται σε διακυβερνητικό διμερές επίπεδο. Λοιπόν, αυτά για τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, τοπικό, περιφερειακό, επιχειρηματικό και τις διεθνείς συμφωνίες. Και επανέρχομαι στο πρώτο σημείο κλείνοντας ότι χρειάζεται ότι ναι μεν θα πρέπει να δούμε τι θετικά έχουν γίνει και ε, θα το μεταφέρουμε αυτό στο Ρίο, θα πρέπει ταυτόχρονα να θέσουμε ερωτηματικά για τις δικές μας προσπάθειες για την πρόθεση της αηφορίας. Και θα πρέπει φυσικά να δούμε και πώς επηρεάζουμε εμείς τον υπόλοιπο κόσμο, τι ίχνη δίνουμε εμείς στον υπόλοιπο κόσμο να μην περιοριστούμε μόνο στην αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα, έστω και αν έχει βελτιωθεί η ποιότητά της, να δούμε όμως και ποιοι είναι άλλοι τρόποι με τους οποίους εμείς με τις ενέργειές μας βοηθάμε ή δεν βοηθάμε την αηφορία σε λιγότερο ευτυχή μέρη του κόσμου. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις εσωτερικές μας συμπεριφορές. Σαν παράδειγμα η δίψα που έχουμε για απεριόριστη για προϊόντα ξυλίας από τα τροπικά δάση για πρώτε ύλες που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτική βιομηχανία οδηγούν πράγματι σε υπερβολές στις ε, χώρες αυτές και δημιουργούν επίσης και ε, βιοκαύσιμα, παραγωγή βιοκαυσίμων σε πολλές από τις υποανάπτυξη χώρες με όρους και τρόπους που δεν είναι σωστοί. Το θέμα λοιπόν του πώς επηρεάζουμε τις χώρες αυτές και μέσω των ειδικών μας συμπεριφορών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Ντερε Κόσμπορ. Η Εκοσόκ. Ήδη εκπονεί μια έκθεση, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μετά τη δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση της ανακοίνωσης από πράσινης Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο φθινόπωρο θα αντιδράσουμε όπως, ε, ξέρουμε το αποτύπωμά μας δεν είναι το ιδανικό και πρέπει να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας να κάνουμε κάτι σε σχέση με τον πλανήτη και στην Ευρώπη και αλλού σε σχέση με τον κόσμο. Λοιπόν, φτάνω στο Σάντορ Φιλεπ από την Ουγγαρία που έχει τώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοινοβούλιο έχετε έναν επίτροπο για τις μελλοντικέ γενναίες που είσαστε εσείς στρεφόμενοι στο μέλλον, προσπαθώντας να συνθέσετε όλες αυτές τις απαντήσεις για αυτές τις προκλήσεις, εξηγήστε μας τα σχετικά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πραγματικά ο συντονιστής ε, για τα θέματα μελλοντικών γενεών στο Κοινοβούλιο μας. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα αυτής της, ε, αυτού του αξιώματος που έχω για τις μελλοντικές ε, γενναίες, για τις μετεξελίξεις σε σχέση με το διεθνές και το εθνικό επίπεδο αν με συγχωρέσετε θα ξεκινήσω με κάποια ε, κοινή λογική θέση που πρέπει να επαναλαμβάνεται σε σχέση με τις ε, εκδηλώσεις μας. Οι κοινωνίες μας ε, οι ίδιες αυταπατώνται αποτύχαμε να αναγνωρίσουμε την επιτάχυνση σε σχέση με κάποια περιβάλλοντα που ε, αντιμετώπισαν κρίσεις και σε σχέση και με το μέλλον μας το κάνουμε αυτό. Γιατί το κάνουμε αυτό διότι φυσικά εδώ υπάρχει το συμφέρον, αντικρουόμενα θέματα συμφερόντων όσον αφορά κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Δυσλειτουργούμε λοιπόν στο, θέμα των νομικών ε, διατάξεων και ε, δυνατοτήτων λειτουργίας. Πρέπει από πλευρά των κυβερνήσεων σε σχέση με το, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη να λαμβάνονται αυτά βέβαια υπόψη ενώ υπάρχει ε, σε διαφορετικό επίπεδο αντικρουόμενη δράση. Αυτό είναι σχιζοφρενικό. Βλέπουμε σε διαφορετικό χρόνο την απέτηση λύσεων. Αν έρθουν γοργά οι λύσεις ε, βλέπουμε σε σχέση με την αξιολόγηση των στόχων της χιλιετίας, ε, σε σχέση με το κυβερνητικό επίπεδο και τις διαφορετικές δράσεις όπως και ανεξάρτητων ε, ε, ερευνητικών οργάνων. Βλέπουμε τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών. Βλέπουμε εναλλακτικές δυνατότητες από τις τοπικές κοινωνίες ε, και ομάδες για τοπικές λύσεις, για ενεργειακά θέματα, θέματα που αφορούν τα, την, τα τα, το, το υδάτινο περιβάλλον κτλ. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία το Ρίο 20 ε, ως ε, εκδήλωση να εισαχθούν κάποιες νέες προτάσεις για λύσεις, διότι το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ή καθορίζοντας ε, την κατεύθυνση σε σχέση με το Ρίο συν 10 έκανε ακριβώς λόγο για αυτά τα προβλήματα και για τις εφικτές πιθανές λύσεις και για αυτά που θα μπορούσαν να είναι η συνεισφορά της Ευρώπης. Εδώ εγώ θα πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει υψηλό επίπεδο πολιτισμού και επιστημονικού παρελθόντος για την αποσαφήνιση αυτής της συστημικής προσέγγισης και αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής και άλλων κρίσεων. Θα μπορούσε να προσφέρει καλά παραθετικά παραδείγματα η ε, Ευρώπη αναφέρθηκαν ε, οι, τα θέματα των, ε, ε, των συμβάσεων που έχουν συναυθεί επαναστατικού χαρακτήρα. Είναι, υπάρχουν λοιπόν διεθνείς συμφωνίες. Δεσμεύονται τα συμβαλόμενα μέρη να αναλάβουν προσπάθειες για θεσμικές λύσεις. Και αυτό είναι πραγματικά η απέτηση των κανονισμών εκείνων που σε συνδυασμό πρέπει να δράσουν με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να δώσει και καλά παραδείγματα η Ευρώπη, όπως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, του Φινλανδικού Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές γενναίες, ε, την Ουγγρική προσέγγιση και άλλες. Ας μιλήσω λοιπόν υπό το πρίσμα του συνηγόρου, του ε, εκπροσώπου ως συντονιστού για τις μελλοντικές γενναίες στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Έχουμε θετικά βιώματα και πείρα όσον αφορά τη δράση μας και θα έλεγα ότι υπό το πλαίσιο αυτού του θεσμού του Ombudsman που επινοήθηκε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της, των συστημικών προβλημάτων που, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συστημικά αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συγκυρία διότι είναι ένα ανεξάρτητο, ένας ανεξάρτητος φορές, ένα ανεξάρτητο σώμα αλλά συντιθέμενο από διαφορετικές τομεακές συνεισφορές με την κατάθεση για παράδειγμα ε, ετοιμάτων ή παραπώνων μπορούμε να δράσουμε και να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες και μη κυβερνητικέ οργανώσεις να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους προβλήματα και μπορούμε να συλλέξουμε αυτά τα βιώματα, αυτή την πείρα και να, θέσουμε, να τα θέσουμε στην ε, ε, υπηρεσία των νομοθετών. Με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να δράσει καλύτερα ο νομοθέτης, το κοινοβούλιο μας. Κάνουμε και ερευνητικό έργο με αυτές τις συνιστώσεις. Βλέπουμε ότι απαιτείται αποσαφήνιση πολλών θεμάτων. Αυτός είναι ο κρίκος που απουσιάζει και πρέπει να συμπληρωθεί. Ας επανέλθω στην ανεξαρτησία μας, στον α, κυρίαρχο ανεξάρτητο χαρακτήρα μας. Είμαστε ανεξάρτητοι και υπό το μεθοδολογικό πρίσμα. Ο Ombudsman λοιπόν για τις μελλοντικέ γενναίες δεν δεσμεύεται με κανένα τρόπο και δεν περιορίζεται με οποιοδήποτε κλάδο της διοίκησης ούτε και με οποιοδήποτε κλάδο επιστημονικό ή άλλο. Είμαστε ανεξάρτητοι και μπορούμε να δράσουμε στο επίπεδο έρευνα, στο ερευνητικό επίπεδο, πολυτομεακά και πολυεπιστημονικά. Είμαστε επίσης ανεξάρτητοι από τις διεργασίες και διαδικασίες και επιβαρύνσεις γραφειοκρατικά ή διοικητικά. Και από πλευράς χρονικής διάστασης μπορούμε να αναλώσουμε χρόνο επαρκή αν αυτό απαιτείται. Και στην διοικητική σφαίρα πραγμάτων και δράσεων τα θέματα των περιβαλλοντικών ε, συνιστοσών δεν μπορούν επαρκώς να καλυφθούν διότι υπάρχει λήψη χρόνου. Είναι μια παγίδα που πρέπει να προσπαθήσουμε πάντα να αποφύγουμε, να αποφεύγουμε. Όσον αφορά τώρα τις μελλοντικές γενναίες για τις δράσεις μας και τα αποτελέσματα, είναι ένα μικρής εμβέλειας γραφείο με λίγους απασχολούμενους δεν μπορούμε παρά μόνο 100 υποθέσεις όσον αφορά το περιβάλλον να αντιμετωπίζουμε αιτήσια, αλλά αυτό έχει σημαντική επίπτωση για τις τοπικές κοινότητες, δήμους, κοινότητες όπως προανέφερα. Και ας επανέλθω στις μεθοδολογικές δράσεις μας α, υπό το θεσμό μας. Προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε το σκηνικό των περιβαλλοντικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Απαιτούμε και συλλέγουμε όλα τα στοιχεία, όχι μόνο από μία αρχή, αλλά από όλους, ώστε να μπορέσουμε και με τις κυβερνητικές, κυβερνητικές οργανώσεις να αντλήσουμε στοιχεία, έχουμε μια διαδραστική προσέγγιση και διεργασία. Συντάσσουμε τα συμπεράσματά μας και τα διανέμουμε και τα διαχέουμε όσον αφορά τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρακολουθούμε με επιτήρηση, εποπτεία στη συνέχεια. Όλα αυτά τι συνεπάγονται. Είναι σημαντικά για τις τοπικές κοινότητες και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Συλλέγουμε όμως και την πείρα και τα βιώματα άλλων και καταλήγουμε σε νομοθετικές προτάσεις που διατυπώνουμε όταν χρειάζεται. Κάνουμε επίση έρευνα όσον αφορά τα κλιματικά, κλιματολογικά θέματα, εναλλακτικέ ε, δράσεις, ε, δείκτε πέρα από το ΑΕΠ, ε, αηφορία όσον αφορά τη δράση των κοινοτήτων μας και το πρασίνισμα του προπολογισμού δημοσιονομικά. Προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές εντάχει όπως θα αναμένατε από μια τέτοια σύντομη εισαγωγή πρέπει να πω ότι προτείνουμε ε, από πλευράς του Ombudsman για τις ε, μελλοντικές γενναίες μέτρα εθνικά, τοπικά και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών που θα μπορούσαν να αναλυθούν υπάρχει πραγματικά διαδεδομένη απογοήτευση όσον αφορά την κρίση, την περιβαλλοντική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να αποσαφινιστούν τα πλαίσια στα οποία κινούμαστε όσον αφορά αυτά τα προβλήματα και να δράσουμε σωστά. Μια, οι δυο μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, όσον αφορά αυτό το πλαίσιο συνοδεύουν και δεν μπορούμε να είμαστε εμείς απομονωμένοι σε ένα σε στεγανό πλαίσιο από άλλους και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και σε τοπικό επίπεδο. Και ε, η Διεθνής Υπηρεσία του θεσμού μας έκανε μια σύντομη ανάλυση και εξι 7 οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών που ήδη έχουν εποπτικές δράσεις, ε, ε, ε, δράσεις εποπτείας για όλα αυτά τα δίκτυα και τις δράσεις συνεπάγονται ένα υψηλό επίπεδο για τις, την διαφύλαξη των συμφερόντων αυτών για τις μελλοντικές γενναίες. Κάτι τέτοιο δεν θα συνεπαγόταν μεγάλες δαπάνες. Έχουμε τις υποδομές. Θα απέστελε ένα πολύ στεναρό ισχυρό μήνυμα προς τους πολίτες για την συνιστόσα για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές δράσεις για το ε, Ρίο 20. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ θερμά. Σάντορ Φίλεπ ένας παγκόσμιος ομπουτσμαν που θα μπορούσε να διοριστεί για την αηφορία των μελλοντικών γενεών. καινοτόμα αυτή η πρόταση που υποβάλλεται. Δίνω τον λόγο τώρα στην συνέχεια στην Μάγια διευθύντρια όσον αφορά την, ε, ε, την Future Justice ε, Department. Και έτσι από πλευρά αυτής της προσέγγισης θα προσδοκούσαμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα και να πω τα εξής. Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την διακυβέρνηση, αλλά και μετά για το τι κάνει το δικό μας ε, Συμβούλιο ε, για το μέλλον. Θεωρούμε ότι ο θεσμό του διαμεσολαβητή είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την ε, εφαρμογή αυτών των αλλαγών. Θα αποτελούσε μια κληρονομιά και για, τον, για τους αστέγους ε, κάτι που αναφέρθηκε στην Υόρκη σε μια πρόσφατη συνάντηση. Δηλαδή, οι άνθρωποι στους δρόμους της Νέας Υόρκης αναφέρονται «Μα τι στο καλό κάνουν αυτοί εκεί στην, ε, στη, στα Ηνωμένα Έθνη». Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάτι και για τους απλούς ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο. Γι' αυτό και ένα τέτοιο θεσμό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συμπληρωματικός ε, ε, κρίκο ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και στα ενδιαφέρομενα μέρη αλλά και για τι κυβερνώσει να συλλέγουν, να φουγκράζονται τις ε, ε, των πολιτών και τα σημεία όπου δεν έχουν σημειωθεί επιτυχίε σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση. Δηλαδή οι πολιτικέ αυτέ είναι θεωρητικά, είναι καταπληκτικές, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Πολύ σύντομα να σα ενημερώσω τι έγινε στην ε, πρώτη ε, διάσκεψη για ε, την αηφόρα ανάπτυξη. Μία διαδικασία μεταβολής από, από το θεωρητικό σχέδιο σε ένα συνεχώς προσαρμοζόμενο πρότυπο. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με πολλές ε, εδρεωμένες ε, ε, πρακτικές. Θα πρέπει λοιπόν να συμφιλιώσουμε τον βραχυπρόθεσμο εκλογικό κύκλο με την μακροπρόθεσμη θέση πολιτικών, τους στόχους οικονομικής ανάπτυξης με την στενή έννοια του όρου, με την ευρύτερη οικονομική και περιβαλλοντική αηφορία. πολύ ε, σημαντική ευκαιρία να ε, έρθουμε σε επαφή με τον πληθυσμό, δηλαδή όχι απλά να τους αναφέρουμε αριθμητικά στοιχεία. Να σκεφτούμε όλοι μαζί την διαδικασία, πώς μπορούμε να τα εξετάσουμε από κοινού και έτσι να τους δείξουμε τις νέες δυνατότητες, τις χρήσεις μετρήσεων για μια νέα διαδικασία ε, και την ενδυνάμωση νέων συμμαχιών μεταξύ ανθρώπων που κανονικά ούτε καν θα μιλούσαν μεταξύ τους. Έχουμε λοιπόν πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες να βελτιωθούμε. Το τρίτο σημείο, ε, σημείο πλεονεκτήματα της ε, συνεκτικότητας και συνοχής ε, των πολιτικών σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης. Θέλουμε να έχουμε μια κοινή βάση λοιπόν στα Ηνωμένα Πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλες τι διάφορες χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς να ε, αναπτύξουν αυτό το κοινό όραμα για, για τον κοινό μας πλανήτη. Και στο πλαίσιο αυτό να βρουν ε, διαφοροποιημένες ε, λύσεις. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το στοιχείο της ε, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Τώρα βλέπουμε ότι η πρόοδος ε, είναι αργή και ε, λόγω και της αποδυνάμωσης του αρμόδιου ε, συμβουλίου ε, επιβραδύνεται ακόμα περισσότερο αυτή η πρόοδος. Το περσινό βαρόμετρο έδειξε ότι 74% των Ευρωπαίων λένε ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση για να καλύψουμε τις ανάγκες του μέλλοντος και 75% συμφωνούν ότι οι πολιτικές πρέπει να προστατεύουν τις μελλοντικές γενιές ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται θυσίες για την τρέχουσα γενιά. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στον ορισμό της ε, αϊ-φόρου ανάπτυξης προκειμένου να διασφαλίσουμε με την ευημερία της τρέχουσας ε, γενιάς χωρίς όμως να διακυβεύουμε το μέλλον, ε, τη ζωή των μελλοντικών γενεών. Ενδεχομένως, τα, οι επιπτώσεις ε, του μη αποδοτικού μοντέλου που ακολουθούμε να είναι τόσο ε, προφανείς στο ευρύ κοινό ε, που δημιουργεί αυτό τέτοια δυσαρέσκεια. Γι' αυτό το ορίο συν έχει αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία ε, να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια με, με πολλά διαφορετικά ενδιαφέρομενα μέρη και με νέες δεσμεύσεις η έκθεση ήδη είχε εντοπίσει αυτή την έλλειψη της ε, συμμετοχής των ε, νέων σε αυτή την δυνατότητα. Και αυτό το κάνουμε, λέει η έκθεση, γιατί μπορούμε. Ε, οι μελλοντικέ γενιές δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τις επιλογές μας. Όμως, ε, οι επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνονται μεταβάλλουν σημαντικά το, τις γενιές αυτών των μελλοντικών γενεών. Αυτό το 1987. Αυτή η μελλοντική γενιά πλέον είναι 23-24 χρονών. Και βεβαίως ε, οι άνθρωποι αυτοί ανησυχούν για την ε, κατάσταση αυτή. Πρώτος σύμμαχός μας λοιπόν για, αυτό το, για αυτή τη διαμεσολάβηση που θα υπάρχει μέσα στο, στα πρώτη διακυβέρνηση είναι αυτή η νέα γενιά. Κατανοούν, ε, επιθυμούν την εξέβρεση λύσεων, έρχονται, ξαναφεύγουν γιατί απογοητεύονται. βλέπουν ότι τίποτα δεν συμβαίνει και πολλοί έχουν την αίσθηση ότι αυτές οι διαβουλεύσεις δεν ε, έχουν κάποιο σημαντικό νόημα. Ουσιαστικά δημιουργούν ένα τελείωτο χαρτομάνι χωρίς ε, αυτά αποτελέσματα. Επομένω, το να έχουμε κάποιον μέσα στην κυβέρνηση ε, από τον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες είναι πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για πολύ κόσμο. Και θα βοηθούσε στην παρακολούθηση της εφαρμογής, ε, στην εποπτεία. Πολύ σημαντική ευκαιρία λοιπόν αυτή που έχουμε μπροστά μας για να αυξήσουμε τη συνεργασία. σήμερα έχουμε αυτή την συνεδρίαση. Το απόγευμα η Επιτροπή στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας έχει μια συνεδρίαση εστιάζοντας στον διαμεσολαβητή συγκεκριμένα για το περιβάλλον και εγώ θα ήθελα να συμμετάσχω να όλοι μόνο σε αυτή τη συζήτηση να δούμε τι συμβαίνει με τα υπάρχοντα συμβούλια αηφόρου ανάπτυξης. Όμως υπάρχουν φήμες, όπως αναφέρθηκε, ότι όλη αυτή η ιδέα για την Ευρωπαϊκή Στατική 2020, για την έξυπνη, περιεκτική και αηφόρο ανάπτυξη. Ε, όμως αυτό ε, προσκολάται στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η οικονομία που θα πρέπει να ε, σχεδιάζεται κατά, κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων χωρίς να ε, καταρρύπτει όμως και να καταστρέφει το, ε, την βάση. Δεν βασίζεται λοιπόν σε τρεις πυλώνες αλλά μία σε, σε, σε ένα νέο υπόβαθρο. Ε, η δήλωση που θα προκύψει από το Ρίο, 2020, από το 20 θα μας επιτρέψει ε, να ε, σχεδιάσουμε την ε, μελλοντική μας πορεία. Αν δούμε και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευημερία του πληθυσμού της Ευρώπης είναι ένας από τους κύριους στόχους. Και μετά βέβαια έχουμε και όλη αυτή τη συζήτηση που θα προκύψει από το πάνελ για την αηφόρα ανάπτυξη. Αυτό το πάνελ δείχνει πώς ε, ε, λειτουργεί αυτός ο θεσμός, Τα ανέφερε και ο συνάδελφος. Έχουμε αυτή την, ε, αυτό το θεσμό του διαμεσολαβητή, του Ombudsman. Υπάρχει ο θεσμός, αν και δεν τον έχουν εφαρμόσει όλες οι χώρες. Αλλά μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε περισσότερες προσπαθίες μας. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κυρία η πολιτική για τις ε, μελλοντικές μέλουσες γενναίες ε, είναι ένα πρόβλημα για μια οικονομία που δεν βλέπει πέρα του τριμήνου. Ε, ασχολούνται οι πολιτικοί μόνο λίγο πριν από τις επόμενες εκλογές. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κάποια θεσμικά όργανα και κάποιες μικιό να κάνουν την προσπάθεια αυτή και να μας θυμίζουν ότι όλοι θα πρέπει να παρουσιάσουμε τις επιδόσεις μας. Λοιπόν, ακούσαμε πολλές ιδέες από το δεύτερο πάνελ. Έχω πάντα βέβαια μία μικρή σύγχυση. Γιατί η ιδέα για ένα ombudsman, ombudsman είναι κάποιος ή κάποιο σώμα το οποίο είναι ανεξάρτητο και μπορεί να εργαστεί με ανεξάρτητο τρόπο. Υπάρχουν και οι γνωστές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, δεν ξέρω κατά πόσον συντονίζονται στα πλαίσια ενός συμβουλίου. Θα αναπτύξουμε τη UNEP, το UNDP. Εν πάση περιπτώσει δύο ερωτήσεις, σύντομες παρακαλώ, όποιος θέλει. Αν και δεν έχει ζητήσει κάποιος να θέσει ερωτήσεις, νομίζω ότι το πρωινό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για μας, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό μας. Λάβαμε σοβαρά υπόψη ότι ακούστηκε και ήταν μια καλή προϋπόθεση για τη δουλειά μας ε, τον, το φθινόπωρο που θα παρουσιάσουμε την, πρότασή μας. Ποιος Πέσβης έχει το λόγο. Ένα σχόλιο λέει ο κ. Σταβάρης για κάτι το οποίο έθεσε ο κ. Όσμπορν. Αναφερόμενο στη Βαζιλία και στα βιοκαύσιμα. Ο τέος πρόεδρος Λούλα μας έλεγε ότι η εθανόλη είναι σαν τη χολεστερόλη. Υπάρχει καλή και κακή. Και στη Βραζιλία λοιπόν έχουμε περισσότερο την καλή. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί χρησιμοποιούμε μόνο ένα μικρό τμήμα των ε, εδαφών μας, 1% μόνο, για την παραγωγή εθανόλης από ζαχαροκάλαμο. Έχουμε την υψηλότερη παραγωγικότητα που μπορούμε να πετύχουμε. 7 προς 1 σε σχέση με το καλαμπόκι δεν απειλείται η παραγωγή τροφίμων και είναι και πάρα πολύ μακριά από, την, από τα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Είναι σαν να λέτε ότι η παραγωγή του κρασιού στη Γαλλία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δάση στην Ρωσία. Σας, σας ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Ξέρετε ότι διεξάγεται εντονότατη συζήτηση για τα βιοκαύσιμα, για την πρωτοβουλία αυτή και το κόστος ε, και σε μια μικρή πύρο σαν την Ευρώπη είμαστε πιο ευαίσθητοι για τις παρενέργειες και τις αρνητικές επιπτώσεις. Ε. Εσείς έχετε πολύ μεγάλη έκταση ως ε, εμβαδόν στη Βραζιλία. Παρακαλώ, τα είπαμε όλα. Άλλος. Η ιδέα του Ombudsman, ε, λέει ο Λαλόντ, είναι μια πολύ καλή ιδέα, θα έλεγα. Τώρα, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον Τζο Λάινεν που ήταν στη Στοχόλμη στο παρελθόν, το ίδιο ερώτημα διατυπώνεται. Κάνουμε, σημειώνουμε πρόοδο ή όχι, ή οπισθοδρομούμε. Τζο, όταν ήμουνα φοιτητή, ο όρος οικολογία δεν βρισκόταν ούτε καν στα λεξικά καθόλου ήταν ανύπαρκτος. Σημειώθηκε τεράστια πρόοδος λοιπόν. Τώρα, αν επαρκεί, αν ακολουθούμε ταχύς ρυθμούς ε, σε αυτή την κατεύθυνση για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, ανοιχτό το ερώτημα. Η κατάσταση στο περιβάλλον δείχνει ότι επιδεινώνονται αφενός τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα και στην Ασία, ξεκινώντας την Αφρική, από την Αφρική. Σε λίγα χρόνια η Αφρική θα έχει περισσότερους κατοίκους η Αφρική από ότι η Ινδία, η Κίνα θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τέτοιου είδους ε, ε, προκλήσεις. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και για τις μελλοντικέ γενναίες θα πρέπει να δούμε τον κύριο ρόλο, διότι μετά την ε, αύξηση αυτή θα έχουμε μια σταθεροποίηση του παγκοσμίου πληθυσμού. Και ίσως αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης. Ευχαριστώ. Ο Ντέρεκ προκλήθηκε από τα βιοκαύσιμα ίσως, από ποιο. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον Βραζιλιάνο πρέσβη διότι ε, έκανα κάποια πρόκληση. Δεν ήθελα να διαχωρίσω καλώς, καλά αρνητικά βιοκαύσιμα. Πολύ καλές επιδόσεις έχει η Βραζιλία και υπάρχει και η ανησυχία ίσως να, μην δίνεται, να δίνεται υπερβολική έμφαση στην ανάπτυξη βιοκαυσίμων όπου θα υπήρχε η δυνατότητα ίσως δημιουργίας προβλημάτων στα τρόφιμα για τα τρόφιμα. Ας δεχτεί λοιπόν αυτή την ε, διαφοροποίηση επί της τοποθέτησής μου ο Βραζιλιάνος πρέσβης σε αυτό που είπα πριν. Ήθελα να προσθέσω ένα πράγμα για την ιδέα του Ombudsman, ενδιαφέρον θέμα που θα έπρεπε να τύχει συνέχεια και να διερευνηθεί. Θα έπρεπε όμως παράλληλα με τις άλλες προτάσεις να διερευνηθεί που δεν αναφέρθηκαν και που από πλευράς των μελών του Ευρωκοινοβουλίου θα έπρεπε να δειχθεί ενδιαφέρον σε αυτό. Δηλαδή να υπάρξει ένα διεθνές, ένας διεθνής περιβαλλοντικός οργανισμός να υποστηρίξει τις, ε, τις κυβερνητικές ε, προτάσεις και ε, ιδέες, ιδέες που υποβάλλονται. Ίσως έτσι θα μπορούσε να υπάρξει άρθρωση μιας σωστής ε, δράσης. Αυτό πρέπει να εξεταστεί πιο σοβαρά. Ευχαριστώ. Πράγματι αυτή η Επιτροπή έκανε μια εκδήλωση πριν από κάποιους μήνες από κοινού με ε, άτομα από την ε, Βενετία και από εκπροσώπους ε, ε, διεθνών φορέων και ζητήσαμε να υπάρξει μια μελέτη που έχει, ε, βρίσκεται επί τραπέζης και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα αρκετά σύντομα στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και να δούμε πόσο επαρκής είμαστε στην ενεργοποίησή μας για να προαχθούν αυτές οι ιδέες. Σας ευχαριστώ όλους σας λοιπόν πολύ εν κατακλείδη. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά. Συλλέξαμε, σημειώσαμε πολλές καλές ιδέες και πολλές προτάσεις και θα πρέπει να προαχθούν από το Κοινοβούλιο να τύχουν συνέχεια. Θα έχουμε μια αντιπροσωπεία που θα αποσταλεί σε αυτή τη διάσκεψη στο Ρίο Συν Θα εμπλακούμε και θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση στο και εμείς. Σας ευχαριστούμε όλους σας. Λίγη συνεδρίασή μας. Ευχαριστούμε και τους Γερμηνείς. Γεια σας.